Euh, Μάλιστα, θα ήθελα καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Προέδρου Γκούσταυσον, Προέδρου της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητος των Φίλων, που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα και μου ζήτησε να προεδρεύσω αυτή την πρώτη ε, ε, σύνοδο της Επιτροπής μας, γιατί αύριο συνεχίζουμε. Σήμερα η εργασία μας εστιάζεται στους στόχους της Βαρκελόνης του 2002 που έλεγε ότι στο σύνολο της Ευρώπης και για να παροτρύνουμε και να προωθήσουμε τη θέση της γυναίκας στη χώρα εργασίας, να έχουμε συστήματα που να επιτρέπουν στο 90% των γυναικών ανάμεσα στα τρία έτη και τη ηλικία υποχρεωτική σπίτι στο σχολείο να βρίσκονται σε βρεφονιπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε ε, να μπορούν και τα παιδιά, τα βρέφη από 0 μέχρι 2,5 ετών να έχουν ε, θέσεις σε βρεφονιδιακούς σταθμούς. Αυτός ο στόχος επετέφθη το 2010 και μαζί με τους εμπειρογνώμονες μας σήμερα το απόγευμα θα ε, εξετάσουμε ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα ενώ βρισκόμαστε ήδη το, στο 2013 ποιες είναι οι χώρες που κατέβαλαν προσπάθειες πώς οι προσπάθειες αυτές ε, ε, έγιναν, ποιος ήταν ο αντίκτυπός τους και μάλιστα αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό γιατί με την κρίση που ξέσπασε από το 2008 υπήρξε πολύ βαρύ αντίκτυπος στη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας και βλέπουμε σαφώς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα είδη φροντίδα των παιδιών παντού, είτε στο αστικό περιβάλλον είτε στο αγροτικό περιβάλλον σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη θέση των γυναικών στην ε, εργασία. Θα ήθελα να χαιρετήσω το σύνολο των επισκεπτών μας που θα παρακολουθήσουν ε, αυτήν την ε, σύνοδο απόψε και ιδιαίτερα την ομάδα του ΣΕΡ που χαιρετίζω σήμερα εδώ και όλος ιδιαίτερος να καλωσορίσω τη συνάδελφο Μαϊκ ε, Κορνέλισεν, η οποία ασχολήθηκε όλος ιδιαίτερος με το θέμα αυτό, ώστε να διοργανωθεί η σημερινή μερίδα εργασίας που είμαι βεβαία ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα με τους ομπειρογνώμονες και για όλα αυτά τα θέματα είτε πρόκειται για θεματικούς εμπειρογνώμονες, είτε για εθνικούς εμπειρογνώμονες. Θα ε, ακούσουμε λοιπόν δύο ομάδες, δύο πάνελ και θα μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων της Βαρκελόνης. Σας δίνω το λόγο λοιπόν κυρία Κορνέλησεν. Yeah, I'll uh, thank you Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στο θέμα της ε, φύλαξης των παιδιών γιατί συνδέεται άμεσα με την οικονομία, με την παιδεία, με την ισότητα των φύλων, ακόμα και με την καταπολέμηση της φτώχειας και βεβαίως και με την ανθρώπινη ευτυχία. Το 2002 στους στόχους της Βαρκελόνης κάναμε κάποιες επιλογές. Έχουν περάσει 10 χρόνια, 10 κράτη πέτυχαν τους στόχους αυτούς, τα υπόλοιπα όχι. Ίσως λοιπόν έφτασε η ώρα να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές και ειδικά σε αυτή τη συγκυρία της κρίσης όπου σε κάποια κράτη είχαμε επαναχωρήσει σε σχέση με την πρόοδο που θα είχαμε θελήσει να επιτύχουμε στις, ε, στη μέρημνα των παιδιών δεν είναι πάντα το ίδιο σημαντική στις χώρες αυτές η φροντίδα ε, των παιδιών και οι σταθμοί ε, οι βρεφονιπιακοί αποτελούν πλέον μια πολυτέλεια ε, η οποία αντίθετα θα έπρεπε να καλύπτεται ως είδος πρώτης ανάγκης. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη για παράδειγμα τα οποία δεν επενδύουν επαρκώς σε τέτοιου είδους σταθμούς και δεν έχουν τα χρήματα για να καταστήσουν τα συστήματα που στείλουν αποτελεσματικά. Ξέρετε πως για να αυξηθεί το ποσοστό της γυναικείας απασχολησιμότητας θα πρέπει να έχουμε περισσότερους σταθμούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς και παιδικούς σταθμούς. Διάβασα κάπου πως αν είχε οργανωθεί σωστά η φύλαξη των παιδιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απασχόληση των γυναικών θα ενισχύεται κατά τουλάχιστον 1%. Καταλαβαίνετε και ε, το φορολογικό έσοδο ε, ποιο θα ήταν ε, για πολλά κράτη. Σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να καλύψει και τις αυξημένες επενδύσεις που χρειάζονται να γίνονται σε κτίρια και πόρους. Ίσως θα μπορούσε να αυξηθεί και το ποσοστό γονιμότητας. Δεν θεωρώ πως αυτό θα πρέπει βεβαίως προσωπικά να αποτελέσει έναν ιδιαίτερο στόχο, αλλά σε κράτη όπως για παράδειγμα η Σλοβακία, όπου η γεννητικότητα είναι πλέον εξαιρετικά χαμηλή, κυρίως στις αποφύτους ε, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί όταν οι γυναίκες δουλεύουν δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους και χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ της εργασίας και των παιδιών. Καταλαβαίνετε πώς είναι τα πράγματα. Προσωπικά δε θεωρώ το φαινόμενο αυτό αποκρουστικό. Ξέρετε πως οι γυναίκες θα γίνουν οικονομικά πιο ανεξάρτητες αν μπορούν και να εργαστούν και να κάνουν παιδιά και με τη σειρά τους αυτό θα μπορούσε να ε, εξαλείψει την φτώχεια γιατί ξέρετε πως ένας μεγάλος ε, παράγοντας που επιτείνει τη φτώχεια είναι οι γυναίκες που χωρίζουν, δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν το βιογραφικό που θα τους επιτρέψει να βρουν δουλειά γιατί έχουν μεγάλα κενά. Ε, πέφτουν λοιπόν στην παγίδα της φτώχειας πολύ πιο εύκολα και αν δεν υπάρχουν οι σταθμοί φύλαξη, χρειάζεται να μένουν στο σπίτι πολλά χρόνια, όσο τα παιδιά τους είναι μικρά τότε λοιπόν είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος να παραμείνουν στη φτώχεια και το ίδιο συμβαίνει και με τις συντάξεις. Πολλές φορές δεν έχουν αρκετό αριθμό ασφα... Ε, ενσύμων ή ικανή ασφαλιστική κάλυψη έτσι ώστε να έχουν μία αξιοπρεπή σύνταξη. Και πολλές φορές η ερώτηση είναι εξής. Πού μπορώ να αφήσω το παιδί μου και να αισθάνομαι ήσυχη. Αυτό το έχω ζήσει και εγώ. Έχω δύο αγοράκια. Το μεγαλύτερο είναι 5,5, το μικρό είναι 2 και αυτή τη στιγμή ακόμα πηγαίνει στο βρυφονιπιακό σταθμό. Έχουν έρθει και στο Βέλγιο σε βρυφονιπιακό σταθμό, έχουν πάει και στην Ολλανδία και πρέπει να σου πω πως σε δύο χώρες τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Στις κάτω χώρες δεν χαίρομαι όταν αφήνω το παιδί μου το πρωί. Συμπαθητικοί είναι βέβαια όσοι τα φροντίζουν, αλλά οι εγκαταστάσεις το μόνο που κάνουν είναι να αλλάζουν πάνω, να το ταΐζουν και να το βάζουν να κοιμηθεί το μεσημέρι. Και οι άλλες μητέρες πιέζουν, ε, πιέζουν η μία την άλλη, γιατί λένε, ας τέσσερις μέρες το στέλνεις το παιδί σου, τρεις είναι το σωστό, τέσσερις είναι ε, υπερβολικό. Ε, εγώ δεν το πηγαίνω καν μόνη μου το παιδί μου, οπότε καταλαβαίνετε τι άποψη έχουν για μένα και δεν τους νοιάζει που έχουν πατέρα στο σπίτι τα φροντίζει. όχι. Η πίεση υπάρχει. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα στις κάτω χώρες. Έχουν ε, μειώσει τα επιδόματα για τη φροντίδα των παιδιών με αποτέλεσμα σε δική μου οικογένεια να θεωρούμε ότι το εισοδηματικό κριτήριο με αποκλείει από επιδότηση για βρεφονιπιακό. Άρα λοιπόν όλος ο μισθός του άντρα μου ε, χρησιμοποιείται για να πληρώσουμε το βρεφονιπιακό. Και βέβαια επειδή ο άντρας μου θέλει να δουλεύει, τον πληρώνουμε. Σε πολλές λοιπόν οικογένειες όπου η μητέρα συνήθως έχει το χαμηλότερο μισθό, πάβει να δουλεύει. Εάν δουλεύει για να πληρώσει μόνο το βρεφονιπιακό σταθμό, ε, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό όμω μειώνει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Η βελγική μου εμπειρία είναι τελείως διαφορετική. Πάντα πήγαινα τα παιδιά μου εδώ στο βρυφονιπικό σταθμό με χαρά. Δεν είναι ότι τα αλλάζουν και τα ταΐζουν και τα κοιμίζουν το μεσημέρι. Τα διδάσκουν, τα μαθαίνουν γράμματα. Κάνουν μια προσπάθεια να προσαρμόσουν τα παιδιά σε μια μαθητική διαδικασία έτσι ώστε να μπουν ομαλά στη μαθητική ζωή. Και υπάρχει και μια κλίμακα εισοδηματική, οπότε αισθάνεσαι ότι και το ποσό που πληρώνεις έχει υπολογιστεί δίκαια. Με ικανοποιεί, είναι χαρούμενα τα παιδιά, και πρέπει να σας πω πως διάβασα πολύ προσεκτικά αυτό το κείμενο το Σαββατοκύριακο με τα αποτελέσματα της έρευνας και επιβεβαιώνει τις σκέψεις μου. Δηλαδή, δείχνει πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη και τελικά, αν ζεις στη Σλοβακία δεν θες να είσαι η οικογένεια με μικρά παιδιά, στη Γερμανία είτε στην Πολωνία, αν δουλεύουν και οι δύο γονείς, γιατί τότε τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα ήθελες να ζεις στο Βέλγιο, στη Δανία και σε άλλα σκανδιναβικά κράτη, γιατί τα πράγματα είναι οργανωμένα πολύ καλύτερα. Αυτό που δεν είχα καταλάβει και το έμαθα από αυτό το κείμενο είναι πως η νοτροπία η οποία οδήγησε στο να έχουμε βρυφονιπιακούς σταθμούς ε, είναι διαφορετική από κράτος σε κράτος. Είναι κομμάτι η βρεφονιπιακή σταθμή του εκπαιδευτικού συστήματος που σημαίνουν για την ανάπτυξη των παιδιών ή είναι απλώς μόνο για να μπορούν οι γυναίκες να δουλεύουν. Και φαίνεται πως ε, γίνονται λιγότερες περικοπές λόγω κρίσης στα κράτη όπου η αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών είναι κομμάτι του παζλ. Στις κάτω χώρες δεν ήταν ποτέ και δεν υπάρχει καμία πραγματική σχέση μεταξύ των βρεφονιπιακών ε, και του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ σύντομη και έντονη διαφοροποίηση για τα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι λιγότερο ικανοποιητικό για σένα να πας τα παιδιά σου στο σταθμό. Η ποιότητα είναι χαμηλότερη. Και για μένα αυτό ήταν ένα καλό δίδαγμα. Νομίζω πως θα πρέπει να διαβάσετε και εσείς ε, αυτό σας συστήνω την έκθεση. Πολλά μπορούν να μάθουν τα κράτη-μέλη αν εξετάσουν την ε, εμπειρία αλλήλων. Πρέπει να επενδύσουμε στους βρυθονιπιακούς και έτσι επενδύουμε και στην αγορά εργασίας γιατί το μεγαλύτερο ενδυνάμει κομμάτι που θα μπορούσε να ενταχθεί στην αγορά εργασίας είναι οι γυναίκες έτσι ώστε να προλάβουμε τη μελλοντική φτώχεια και έτσι επενδύουμε και στις οικογένειες έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν επιλογή, να κάνουν παιδιά ή να μην κάνουν και να μην εξαρτώνται και να μην χρειάζεται να νομίζουν ότι πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της δουλειάς και των παιδιών. Και σίγουρα είναι και μία επένδυση στα ίδια τα παιδιά. Γιατί στις χώρες όπου αυτή η φροντίδα ε, θεωρείται ως κομμάτι της αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής τους ε, διαδικασίας. Η ποιότητα είναι πιο ψηλή και δεν κινδυνεύουν οι σταθμοί από περικοπές. Νομίζω πως είμαστε στην κατάλληλη στιγμή για να ξαναδούμε τους στόχους της Βαρκελόνης. Και ελπίζω πως μετά το εργαστήριό μας θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και ενδεχομένως να θέσει ένα νέο κεφάλαιο με νέους στόχους για τα επόμενα χρόνια το Συμβούλιο. Merci. Euh. Σας ευχαριστώ, κυρία Κορνέλησεν. Βρίσκω πως πολύ καλά θέσατε το θέμα με συγκεκριμένα και ζωντανά παραδείγματα και βλέπουμε σαφώς τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παρουσία των γυναικών στο χώρο εργασίας και τους τρόπους φροντίδας των παιδιών. Πιστεύω πως επίσης πρέπει να διευρυνθεί αυτό το πεδίο αναλύσεως βλέποντας πόσο πολύ τα είδη φροντίδας επιτρέπουν ισότητα γυναικών ανδρών στην εργασία, στο μισθό αλλά και στη σταδιοδρομία. Και έπειτα το είπατε, είναι ένα στοιχείο φτώχες το να μην υπάρχουν τρόποι φροντίδας ε, του παιδιού για να, και να αναγκάζονται οι γυναίκες να πάψουν να εργάζονται. Αλλά και αυτή η φτώχεια δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να σωρεύεται στη διάρκεια των ετών και τελικά καταλήγουμε με γυναίκες στη σύνταξη εξαιρετικά φτωχές. Μεγάλη δηλαδή απόσταση ανάμεσα στην σημασία των πολιτικών παιδείας και κατάρτισης και στη συνέχεια τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν για να υπάρχει αυτή η πραγματική ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες στο χώρο εργασίας. Θα δουλέψουμε λοιπόν σε ένα πρώτο πάνελ με την Μουριέλ ε, Μπισιέχα της ε, Μονάδας ε, για την Ισότητα των Φύλων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κατή Μακράκεν από το Ίδρυμα Opsit Research του Λονδίνου και την κυρία Πλαντέγκα που έρχεται από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, το τμήμα οικονομικών μας παρουσιάσει το έγγραφο η κυρία Μπισιέρ ε, που παρουσιάστηκε το περασμένο Ιούνιο. Ε, αυτό το έγγραφο αξιολογεί τις προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά τη δημιουργία υπηρεσιών υποδοχής ε, και φροντίδας των παιδιών στην Ευρώπη στα διάφορα κράτη. Δεν θα προσεγγίσει δε μόνο τα εμπόδια και τι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα κρατη να απτύξουν αυτές τις υπηρεσίες για τα βρέφη και τα νήπια, αλλά θα μας ε, επιβεβαιώσει και τους στόχους της Βαρκελόνης, θα μας αποδείξει πως η Κομισιόν ε, δεσμεύεται να στηρίξει τα κρατημέλη ώστε να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους, διότι πίσω από αυτούς τους στόχους υπάρχει και ο στόχος της Ευρώπης 2020 για την πρόθεση της ισότητας των φύλων και την ανάπτυξη της απασχόλησης. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα σας παρουσιάσω την κατάσταση προόδου όσον αφορά την επίτευξη στόχων της Βαρκελόνης. Το πλαίσιο ήδη σας παρουσιάστηκε πολύ καλά. Θα σας δώσω λοιπόν μια εικόνα, την εικόνα μάλλον, και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο ορισμός αυτών των στόχων λοιπόν αναφέρθηκε και σας θυμήθηκε. Να θυμίσω ότι την αρχική σύνοδο το 2010, όπου τα κράτη-μέλη επανέλαβαν αυτά στους στόχους για την του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και έφεραν τη νέα προθεσμία ε, στο 2020. Γιατί να επιτευχθούν οι στόχοι της Βαρκελόνης. Η κυρία Κορνέλησεν ανέφερε γιατί ήταν σημαντική και πώς συνέβαλαν, ε, βρίσκονται μάλλον στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών και συμβάλλουν στην επίτευξη σπουδαίων στόχων όπως η στρατηγική 2020 για τα θέματα απασχόλησης, για τα θέματα εκατάρρησης της και για τη μείωση της εγκατάλειψης των σπουδών. Αυτό επίση είναι σημαντικό για την επίτευξη των στόχων ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και ήθελα να σας θυμίσω δύο γραφήματα για να σας το αποδείξω αυτό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην απασχόληση των μητέρων με μικρό παιδί και τη συμμετοχή των παιδιών στις δομές φροντίδας και βλέπουμε πως υπάρχει μια αρκετά έντονη σχέση ανάμεσα στα δύο. Ένα δεύτερο γράφημα σας δείχνει τη σχέση ανάμεσα στην παρουσία των παιδιών στις υπηρεσίες φροντίδας και το κενό στην αμοιβή ανάλογα με το φύλλο. Όταν δηλαδή η παρουσία είναι, των παιδιών στη φροντίδα είναι υψηλή, τότε μικραίνει το κενό, η διαφορά μισθών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Θα σας δείξω τώρα μια κατάσταση πρόοδου. Αυτή η διαφάνεια δείχνει μια ε, φωτογραφία που αφορά την επίτευξη των στόχων το 2011. Βλέπουμε τρεις ομάδες χωρών. Στο πράσινο βλέπουμε τις έξι χώρες που έχουν επιτύχει τους δύο στόχους το 2011. Στην κρή ομάδα βλέπουμε τις χώρες που έχουν επιτύχει έναν από τους στόχους. Δεξιά από τον ε, κάθετο άξονα υπάρχουν αυτές που έχουν επιτύχει το στόχο για τα πιο μικρά παιδιά και πάνω από τον ορίζοντιο άξονα αυτούς που το πέτυχαν για τα πιο μεγάλα παιδιά. Μετά στην ομάδα την Πορτοκαλί έχουμε χώρες που κοντεύουν να φτάσουν το στόχο, δηλαδή κατά 25% για τα μικρά παιδιά και 80% για τα πιο μεγάλα παιδιά και έχουμε και μια ομάδα που δυστυχώς είναι αρκετά μεγάλη ακόμα και είναι τα κρατημέλη που πρέπει ακόμα να κάνουν σημαντικές προσπάθειες για να επιτύχουν τους δυο στόχους. Τώρα, εδώ πιο συγκεκριμένα έχουμε την κατάσταση προόδου για τα παιδιά 0 με 3 έτη. Οι στήλε αντιπροσωπεύουν τα στοιχεία για το 2010 και τα μικρά κόκκινα σημάδια είναι τα στοιχεία για το 2011. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2010 και το 2011 έχουμε 10 χώρες που έχουν επιτύχει αυτό το πρώτο στόχο. Βλέπουμε επίσης εδώ ότι το ποσοστό παρουσία στις υπηρεσίες διαφέρει. Ας πούμε, με πορτοκαλί έχουμε τις υπηρεσίες τις οποίες ε, πηγαίνουν τα παιδιά για λιγότερο από 29 ώρες την εβδομάδα και στο πράσινο αυτές ε, που τα παιδιά πηγαίνουν για πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα. Ακόμα και αν έχει επιτευχθεί ο στόχος, ε, βασικά είναι μερικοί η επίτευξη όπως της κατοχώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτό το γράφημα λοιπόν βλέπουμε χώρες όπως η Τσεχία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία που βρίσκονται κάτω από το 5%. Εδώ βλέπουμε ε, ότι το 2010 είχαμε ακόμα 10 χώρες που είχαν επιτύχει το στόχο, αλλά το 2011 έχουν μείνει μόνο 9, διότι υπήρξε μια επιστοδρόμηση κυρίως για την Ιρλανδία και την Ισπανία. Για τις κάτω χώρες είναι πάλι επιστοδρόμηση αλλά σε λιγότερο βαθμό. Αντίθετα η Ιταλία προχώρησε. Παρατηρούμε ακόμα ότι η Πολωνία και η Ουγγαρία βρίσκονται κάτω από το 25% της επίτευξης του στόχου. Alors, euh, Ποιοι είναι οι φραγμοί, ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν οι γονεί και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίε. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι το 25% των μητέρων που είτε δεν εργάζονται είτε εργάζονται μερικώς για λόγους ε, φροντίδας των παιδιών, οι δυσκολίες συνδέονται με την διαθεσιμότητα ε, τέτοιων υπηρεσιών. Για τις 53%, το κόστος είναι το πρώτο εμπόδιο και η ποιότητα ακολουθεί. Μόνο στο 4% των περιπτώσεων είναι εμπόδιο και σε 18% των περιπτώσεων υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης. Και τι εννοούμε εδώ. Είτε η απόσταση χιλιομετρική, είτε ώρες ε, ε, λειτουργίας που δεν είναι κατάλληλες είτε ακόμα ε, κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία μπορεί να είναι πολύ περιοριστικά. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως το κόστος παραμένει το βασικό εμπόδιο για τις περισσότερους γονείς. Εδώ τώρα σε αυτό το γράφημα βλέπουμε πως το κόστος είναι ψηλό, αλλά συνήθως αντισταθμίζεται από επιδόματα ή άλλου είδους επιδοτήσεις. Ωστόσο, παραμένει ψηλό το βλέπουμε ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ιρλανδία που το κόστος αντιπροσωπεύει πάνω από το 41% του καθαρών εισοδημάτων σε ένα νοικοκυριό όπου οι δύο γονείς εργάζονται. Επίση, ε, το κόστος των υπηρεσιών θα πρέπει να σχετιστεί και με το κόστος άλλων πολιτικών κοινωνικών ή φορολογικών που επηρεάζουν το εισόδημα μια οικογένεια. Γιατί ακόμα και όταν επιδοτείται εντόνω το σύστημα μέρημνα των παιδιών, Ο δεύτερος γονέας μπορεί να μην συμφέρει να εργάζεται αν φορολογείται υπερβολικά. Το κόστος ε, των υπηρεσιών υποδοχής δεν είναι, επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο τα νοικοκυριά ψηλών εισοδημάτων ή χαμηλών εισοδημάτων. Σε αυτό εδώ το γράφημα μπορούμε να δούμε ότι για τη Γαλλία που είναι άκρια αριστερά ε, θα δείτε πως η μικρή τελίτσα σημαίνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες μέρημνας για τα εισοδήματα για τα νοικοκυριά μάλλον του πρώτου κομματιού εισοδημάτων, του, πρώτου, χαμηλότερων εισοδημάτων και η πάνω βουλίτσα τα ανώτερα εισοδήματα. Η ανισότητα είναι μεγάλη. Ενώ για τη Δανία που είναι δεξιά-δεξιά στο γράφημα, εκεί βλέπουμε πως η κατανομή είναι περίπου η ίδια για όλα τα νοικοκυριά. Δύο λόγια τώρα για την ποιότητα. Είναι πολύ ε, ε, σημαντικό να κάνουμε διάκριση εδώ, να δούμε δηλαδή ε, τα στοιχεία αν είναι συγκρίσιμα, αλλά είναι σημαντικό να δούμε ότι στον τομέα αυτό πολλά παιδιά, πολλοί κόσμος που δεν είναι ιδιαίτερα καταρτισμένος εργάζεται και, το επίπεδο κατάρτισης ή σπουδών είναι πολύ διαφορετικό, είναι επισφαλείς θέσεις εργασίας, είναι ατυπικές, ατυπικά και συμβάσεις ή ε, μερικές. Και δεδομένης αυτής της κατάστασης βλέπουμε ότι οι γονείς χρειάζεται να συνδυάζουν διάφορες λύσεις. Ε, τείνουν να καταφεύγουν στην άτυπη φροντίδα των παιδιών που βασικά εξασφαλίζεται από τους παππούδες και για τις δύο κατηγορίες τις ηλικιακές. Αλλά είναι μερική η φροντίδα, δεν μπορεί, δεν, δεν καλύπτει όλες τις ώρες και άρα χρησιμοποιούνται εναλλακτικές στρατηγικές για να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά. Ε, σε ορισμένε χώρε, λοιπόν το ότι τα παιδιά δεν πάνε στου σταθμού ε, δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ότι ε, δεν υπάρχουν θέσεις. Πολλέ φορέ μπορεί να δίνεται μια ετήσια άδεια για να γονείς στο σπίτι και να φροντίζουν για το παιδί τους ε, για ένα έτος, ε, στο τέλος του οποίου έχουν το δικαίωμα να πάνε το παιδί τους σε κάποιο σε κάποια άλλη δομή, αλλά σε άλλες χώρες υπάρχει ε, πρόβλημα όσον αφορά τις θέσεις φροντίδας των παιδιών και αυτό ε, επιβαρύνει την θέση της γυναίκας στον χώρο εργασίας. Πέρα λοιπόν από τις ποιοτικέ παροχές και σε συνδυασμό με τις γονικές άδειες θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να παίρνει οικογενειακή άδεια και ο πατέρας των παιδιών. Και εδώ έρχομαι τώρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο Αυτό που είναι απαραίτητο είναι μια σφαιρική προσέγγιση που να συνδυάζει ποιοτικές υπηρεσίες υποδοχής, προσιτές, με συστήματα οικογενειακών αδειών που να είναι προσαρμοσμένες, με ελαστικό ωράριο και όλα αυτά κάθε φορά, σε κάθε στάδιο της ζωής, δηλαδή όσο είναι μικρά τα παιδιά, αλλά και όταν πηγαίνουν πια δημοτικό και πέρα από τα σχολικά ωράρια, αλλά και για τους υπόλοιπους εξαρτώμενους της κάθε οικογένειας. Τα φορολογικά εμπόδια αλλά και τα άλλα εμπόδια για την απασχόληση των γυναικών θα πρέπει να καταργηθούν για να μπορεί και, και να μπορεί μάλιστα και ο πατέρας να αναλάβει περισσότερες οικογενειακές ευθύνες. Πρέπει να γίνουν πολλές δράσεις για να προωθηθεί αυτός ο συνδυασμός μέτρων για τον συνδυασμό οικογενειακής με εργασιακή ζωή και η Κομισιόν φυσικά θα συνεχίσει την επιδίωξη και την, για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελόνης. Τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει και στατιστικές δυνατότητες γιατί φαίνεται σημαντικό να έχουμε περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τους φραγμούς την πρόσβαση των υπηρεσιών αυτών. Βεβαίως ε, και η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να στηρίζει ε, αυτές τις προσπάθειες στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, υιοθετώντα συγκεκριμένες συστάσεις και καλώντας τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν τους στόχους της Βαρκελόνης και να διατηρήσουν μια ε, δημόσια επένδυση στον τομέα αυτό παρά την κρίση. Θα καλέσει επίσης τα κράτη-μέλη να εκμεταλλευτούν ε, στο maximum τα διαφορετικά ταμεία. Και εδώ έχετε διάφορες δράσεις, μελέτες που γίνονται για το θέμα αυτό, ανταλλαγές ε, των ε, καλών πρακτικών, αλλά μέσα σε όλα αυτά θα ήθελα να φέρω μια συγκεκριμένη δράση που είναι σημαντική για και σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα της υποδοχής και της φροντίδας των μικρών παιδιών. Μέσα στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού έχει δημιουργηθεί μια θεματική ομάδα εργασίας ε, πολιτικών ηθινόντων, ακαδημαϊκών αλλά και εργαζόμενων στον τομέα ώστε να φτιάξει αυτό το πλαίσιο που θα βασίζεται σε πέντε πτυχές ε, πρόσβαση, συνθήκες εργασίας, ποιότητας, παρακολούθηση και αξιολόγηση, διακυβέρνηση και χρηματοδότηση και έτσι θα έχουμε ένα πρώτο κείμενο τον Ιούνιο του 2014. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω τον τίτλο αυτού του εργαστηρίου, η αναθεώρηση οι στόχοι της Βαρκελόνας ξαναχτυπούν. Νομίζω πως ε, ε, το έγγραφο της Κομισιόν είναι περιστατωμένο. Ε, τονίζεται η σημασία των υπηρεσιών φροντίδας ε, των ε, παιδιών και θα πρέπει αυτό να υποστηριχτεί από τα κράτη-μέλη στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπισιέρ, και το λόγο θα πάρει η δεύτερη εμπειρογνώμων μας, η κυρία Κάθη Μακκράκεν που είναι συντονίστρια από το 2006 ε, μιας ομάδας συμβούλων του Opsit Research. Έχει κάνει ερευνητικές εργασίες και εξεργασίες αξιολόγησης για την Βρετανική κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και για το Ευρωκοινοβούλιο. Προσφάτως μάλιστα έκανε μια έρευνα μετά από αίτημα της Επιτροπής μας που φέρει τον τίτλο «Οι επιπτώσεις της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης στα συστήματα προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας» και πιο συγκεκριμένα θα μας παρουσιάσει σήμερα τα συμπεράσματά της όσον αφορά τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητος στις δομές υποδοχής των νέων παιδιών και την αντίστοιχη κατάσταση των γυναικών και των ανδρών στον χώρο εργασίας. Κυρία Μακράκεν, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε λοιπόν τις ε, πτυχές της κρίσης όσον αφορά τα δύο και τις επιπτώσεις ε, της κρίσης σε γενικότερο επίπεδο. Φυσικά η φροντίδα φροντίδε παιδική μερίμνα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω τα κυριότερα συμπεράσματα της ανάλυσης μας. Η έρευνα είχε να κάνει με μελέτη βιβλιογραφίας, με ανάλυση δεδομένων που είχαμε στη διάθεσή μας, καθώς και με μελέτες περιπτώσεων από κράτος μέλους. Κράτος μέλους. Η κατάσταση πριν την κρίση είχε ως εξής, συνοψίζοντας, τις δύο δεκαετίες ε, που προηγήθηκαν της κρίσης, αυξήθηκαν ε, τα εισοδήματα κατά μέσο όρο σε κάθε χώρα του ΩΣΑ και οι κυβερνήσεις ε, στην Ευρώπη έτειναν ε, στο να αναπτύξουν την οικογενειακή τους ε, πολιτική. Φυσικά η αύξηση του πληθυσμού και γύρανση του πληθυσμού επιβάρυνε πάρα πολύ την ε, πολιτική αυτή και τον περιπολογισμό. Τώρα, να σας πω ότι μιλώντας για υπηρεσίες παιδικής φροντίδας εννοούμε τις επίσημες υπηρεσίες και τα μέτρα ζήτησης και προσφοράς, καθώς και την πολιτική με, για την γονική άδεια, πολιτική φροντίδα των παιδιών κτλ. Μετά το 2008, από τότε που άρχισε η κρίση, ξέρουμε ότι επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση πολλών οικογενειών εξαιτία της ανεργίας τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών. Η απάντηση των ε, κρατών μελών διέφερε. Και αυτό εξαρτήθηκε από το είδος του κράτους προνοίας που υπήρχε σε κάθε κράτος μέλος. Βλέπουμε λοιπόν ορισμένες ε, περιπτώσεις όπου επεκτάθηκε το κράτος πρόνοιας και η οικογενειακή πολιτική συμπεριέλαβε διάφορα μέτρα τόνωσης ε, της ε, οικονομίας ή προσωρινά είτε μόνιμα. Για παράδειγμα, αυξήσεις ε, επιδομάτων, μέτρα έκτακτα, μέτρα αντιμετώπισης κρίσης ή ορισμένα επαναξιολόγηση ορισμένων επιδομάτων. Είδαμε λοιπόν ταυτόχρονα και αυξήσεις των δαπανών και περικοπές των δαπανών. Σημαντικό είναι να δούμε επίσης πώς αντιμετώπισαν ε, την αλλαγή αυτή της οικονομικής τους ε, κατάστασης οι διαφορές οικογένειες ε, και πόσο αυτό επηρέασε τις ώρες εργασίας ανδρών και γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις υπηρεσίες παιδικής μέρημνας ε, σε το γενικότερο πλαίσιο των άλλων υπηρεσιών επρόνοιας. Η απάντηση λοιπόν ε, του κράτου επρόνοια ήταν άμεσα συνδεδεμένη με διάφορους σταθεροποιήτε, για παράδειγμα επιδόματα ανεργίας, τα οποία ενεργοποιούνταν άμεσα από τη στιγμή που κάποιος ε, έχανε την δουλειά του. Έχει αναφερθεί βέβαια ότι οι πρακτικές αυτές πολλές φορές έχουν οδηγήσει σε ανισότητες και σε αύξηση των ανισοτήτων αυτών εις βάρος των γυναικών. Τώρα, αν δούμε τις ε, δαπάνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δούμε ότι οι δαπάνες όσον αφορά τους αυτόματους σταθεροποιητές ε, έτειναν προς αύξηση. Για παράδειγμα, τα επιδόματα παιδιών. Επίσης, οι αυτόματοι αυτοί οι σταθεροποιητές ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με τα επαγγελματικά προσόντα και αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης των γυναικών με λίγα επαγγελματικά προσόντα και λίγες δεξιότητες. Επίσης, άλλα μέτρα αντιμετώπισης σε περίοδο κρίσεως είχαν να κάνουν με διάφορες πολιτικές ανεργοποίησεις εργατικού δυναμικού. Και το ενδιαφέρον με αυτό είναι ότι το κόστος της παιδικής μέρημνας συμπεριλήφθη στο όλο πακέτο αντιμετώπισης. Επίσης, παρατηρήσαμε μία τάση αναθεώρησης του ρόλου του φροντιστή των παιδιών. Είδαμε δηλαδή ότι οι περικοπές που έγιναν οδήγησαν σε μία τάση οι μητέρες και οι γιαγιάδες να αναλάβουν τη φύλαξη των παιδιών, κάτι που στο παρελθόν είχε μειωθεί. Διότι πάρα πολλές το να επιστρέψει μια γυναίκα στο χώρο εργασία ε, σήμαινε και αύξηση των δαπανών. Τώρα Α δούμε τις περιπτώσεις από χώρα σε χώρα. Ελλάδα. Να σας πω ότι κοιτάξαμε τα διάφορα καθεστώτα ε, προνοίας στις ε, διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα λοιπόν Όσον αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης κρίσης, είδαμε μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις και σε περικοπές. Η επίσημη κοινωνική προστασία μετατέθηκε στις οικογενειακές δομές. Με άλλα λόγια, η οικογένεια ήταν εκείνη που παραδοσιακά παρήχε φροντίδα παιδιών. Τώρα, ε, ορισμένες ε, παροχές και ορισμένα επιδόματα είχαν πολύ πιο αυστηρά κριτήρια παροχής. Υπήρξαν επίσης πολλές περικοπές των επιδομάτων που αφορούσαν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες. Περικοπές παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα στις ε, ανήπαντρες μητέρες. Και κάτι παρόμοιο Να μπορείτε να μιλάτε, να, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Στην Ιταλία. Υπήρχε ανέκαθεν μία ανάγκη μεταρρύθμισης του κράτους ε, πρόνοιας, ιδιαίτερα στον τομέα των συντάξεων που επιβαρύνουν το κράτος πρόνοιας. Χρειάστηκε λοιπόν μία αναδιάρθρωση. Έγιναν λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές ε, περικοπές τόσο στις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών όσο και στις υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων. Στην Ιταλία παραδοσιακά οι μεγαλύτερε ηλικίε ήταν αυτέ που αναλάμβαναν την φύλαξη παιδιών. Στην Πολωνία τώρα τα αποτελέσματα και επιπτώσει τη κρίση ήταν λιγότερο αισθητά στον τομέα της ε, παιδικής εμέρημνας. Είδαμε σε γενικές γραμμές ε, μια γενικότερη μείωση των ε, οικογενειακών επιδομάτων, η οποία φυσικά έπληξε περισσότερο γυναίκες. Στη Σουηδία τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Ο δίκτυπος της κρίσης μια συνεχιζόμενη κρίση, έγινε λιγότερο αισθητό στην σουηδική οικονομία. Το σουηδικό μοντέλο, όπω γνωρίζετε, συμπεριλαμβάνει ε, ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων και για τις μητέρε και για τους πατέρε, αλλά και ολοκληρωμένε παροχέ παιδικής μέρημνα από το κράτος οι οποίε βασίζονται σε ένα πακέτο ισότητας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιήθηκε, τέθηκε σε εφαρμογή ένα πολύ αυστηρό σχέδιο λιτότητας και περικοπών. Αυτές οι περικοπές οδήγησαν στη, στη μειωμένη δυνατότητα των ορισμένων οικογενειών να πληρώσουν τις υπηρεσίες ε, παιδικής μέρημνας και αυτό οδήγησε σε πολλά προβλήματα και σε αύξηση του κόστους για βρεφονιπιακό σταθμό. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα συμπεράσματα της έρευνάς μας είχαν ως εξής. Η εισαγωγή πολιτικών ενεργοποίησης του εργατικού δυναμικού ενδεχομένως έχουν κάποιο όφελος για τις γυναίκες. Αλλά εάν δεν δοθεί ιδέουσα προσοχή στις ε, ανάγκες παιδικής εμέριμνας, δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά τις γυναίκες. Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Επίσης, ή περικοπές στις μεσογειακές χώρες και στην Ιρλανδία δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα κονδύλια που περικόπησαν δεν δόθηκαν σε νέες επενδύσεις. Οι συστάσεις μας λοιπόν θα ήταν οι κυβερνητικοί εταίροι να διασφαλίσουν ότι θα διεξάγεται μία ε, ενδελεχής ε, αξιολόγηση αντικτύπου που θα συμπεριλαμβάνει και τις επιπτώσεις των περικοπών στις ε, υπηρεσίες παιδικής μέρημνας χρειάζεται μία εκ νέου εξισορρόπηση των ε, δαπανών. Οι περικοπές δηλαδή που γίνονται σε έναν τομέα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως επενδύσεις για έναν άλλον τομέα. Επίσης χρειάζεται μεταρρύθμιση των διατάξεων όσον αφορά τις αγωνικές άδειες. Merci beaucoup, euh, madame. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μακράκεν για αυτή τη ματιά που ρίξατε η οποία ήταν και σφαιρική. Μας εξηγήσατε πως έχει η κατάσταση με τους βρεφονιπιακούς σταθμού γενικότερα αλλά και πολύ στοχευμένη συνάμα μια και μας μιλήσατε για κάποια, για αρκετά κράτη δίνοντάς μας πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία με πολλές λεπτομέρειες. Θα περάσουμε τώρα στην τελευταία εμπειρογνώμονα στο πάνελ αυτό, την κυρία Γιάννη και καθηγήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σουρτρέχτης. Η έρευνα που κάνει στοχεύει στην ευελιξία της αγοράς εργασίας και στην συμφιλίωση της ιδιωτικής και της εργασιακής ζωής και πιο συγκεκριμένα στην ε, κοινωνική πολιτική που ακολουθείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό ε, επίπεδο. Μιλήσατε για την ανακαδιανομή της μη πληρωμένης εργασίας, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό τώρα στην κρίση, για την αλλαγή των ωραρίων εργασίας στους βρεφονιπιακούς σταθμούς όπως επίσης και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Θα παρουσιαστείτε λοιπόν σήμερα και στα δύο σεμινάρια που κάνουμε. Θα δείχνουμε τη χαρά να σας ακούσουμε δύο φορές και θα μιλήσετε τώρα πρώτα για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή. Ένα θέμα για το οποίο θα σας ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια για, το, για τις ε, εγκαταστάσεις ε, φύλαξης και φροντίδας ε, πολύ μικρών παιδιών που βρίσκονται στον πυρήνα του όλου θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ θερμά για τις προσπάθειες αυτές που κάνετε. is ook vooral in combinatie met Engelse slides. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ehm, Όμως, έχω σημειώσει σε στα αγγλικά, θα μιλήσω Ολλανδικά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να μιλήσω λοιπόν για το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε οικογένεια, παιδιά και εργασία. Ως επιστήμον και ερευνήτρια ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το ότι στην Ευρώπη έχουμε ένα μοντέλο το οποίο μια Βρετανίδα κοινωνιολόγος η Τζέιν Lewis περιέγραψε ως ε, μοντέλο ενήλικου εργαζόμενου. Με γονική άδεια, κοινωνική ασφάλιση, φορολόγηση, μέρημνα παιδιών. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ε, διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Και αυτό αρχίζει από το μοντέλο απασχόλησης, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ενήλικοι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, μπορούν να έχουν δουλειά. Αυτό φυσικά έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στην ε, κοινωνική ατζέντα. Το πόσο μπορούμε να συνδέσουμε την ε, επαγγελματική ζωή με την φροντίδα των παιδιών έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η παραδοσιακή, το παραδοσιακό μοντέλο πολιτικής, ε, τα επιδόματα για τα παιδιά, αγωνικά επιδόματα... οι παροχές αυτές εστιάζονται κυρίως στη φύλαξη των παιδιών και στην γονική άδεια. Όμως αν δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη ιδιαίτερα όσον αφορά το ε, μοντέλο απασχόλησης που έχουμε και την ε, κοινωνική ατζέντα, θα δούμε ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έχουν αντιδράσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παιδική μέρημνα. Η πρώτη ομιλήτρια ήδη έκανα μια πολύ καλή παρουσίαση και θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτά που είπε ότι να προσθέσω ποιε είναι οι μεγάλες ε, διαφορές. Καταρχά, όσον αφορά τι επενδύσει ε, στην παιδική μέρινα. Βλέπετε εδώ τι διακυμάνσει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. 72% στην Δανία, 72% των παιδιών δηλαδή βρίσκονται σε κάποιο βρεφονιπιακό σταθμό ένα ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο. Η πρόκληση λοιπόν στον κλάδο αυτό είναι η διαφορές και η εξισορρόπηση των διαφορών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τρία κράτη-μέλη στα οποία διασφαλίζονται 30 τουλάχιστον ώρες ε, παιδικής εμέριμνας η Δανία, η Σλοβακία και η Πορτογαλία. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει καθεστώ ήμη απασχόληση στην ε, φροντίδα των παιδιών. Επίσης κάποιοι κάτι όπως οι κάτω χώρες έχουν μόνο το 6% των παιδιών τους σε βρεφονιπιακούς σταθμού σε 30 ώρες την εβδομάδα. Η υπόλοιπη, η συντριπτική πλειοψηφία προτιμά την ήμια απασχόληση. Αυτό λοιπόν μας δείχνει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν όσον αφορά τις ε, ώρες φύλαξης ανά εβδομάδα. Βλέπουμε λοιπόν ευθύς εξ αρχής ότι η πλήρης ε, απασχόληση είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η άτυπη παιδική μερίμνα είναι κάτι που παρατηρείται ε, πολύ συχνά. Κάτι δηλαδή που είναι οργανωμένο όχι από το κράτος ή από το δημόσιο. Παιδιά τα οποία φιλάνε συγγενείς ή φίλοι. Εδώ στη δεύτερη στήλη βλέπετε ότι το 50% της ε, παιδικής ε, μέρημνας ε, στην Ολλανδία παρέχεται από κρατικούς φορείς και το 50% από ιδιωτικούς φορείς. Βλέπουμε τις χώρες οι οποίες παρέχουν εξίσου κρατικές και μη κρατικές και άτυπες υπηρεσίες φύλαξης. Να σας δώσω λοιπόν κάποια παραδείγματα. Ιταλία, Κύπρος και Ελλάδα. Εδώ μιλάμε για τα κράτη-μέλη από τον Νότο, όπου ακριβώς ισχύει αυτό. Και χαμηλό, χαμηλές επιδόσεις για την επίσημη ε, φροντίδα και έχουν ε, και χαμηλές επιδόσεις στην άτυπη φροντίδα, ε, τα έχουμε σημειωμένα εδώ. Τώρα, τέλος, εάν θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά γενικότερα, όταν κοιτάζει κανείς την κατάσταση με τα μεγαλύτερης ηλικία παιδιά, δηλαδή τρία ως και την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης, θα δείτε πως οι διαφορές είναι μικρότερες και αυτό σχετίζεται με το ότι οι Αυτές οι ομάδες οι ηλικιακές, ή προσχολικές, ε, καλύπτονται και από κάποιες άλλες ρυθμίσεις ε, απασχόλησης παιδιών. Άρα λοιπόν έχουμε τα όρια μεταξύ βρεφονιπιακού, προσχολικού, προνηπίου, νηπίου, ε, πρώτης δημοτικού με κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες χώρες έχουν η Δανία, για παράδειγμα, ε, προσφέρουν, όπως και η Εστονία και η Σλοβενία, ε, μια κάλυψη 100% του χρόνου και υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, επενδύσει σε δομές μερικής απασχόλησης των παιδιών, όπου μπορεί κανείς να τα αφήσει για ένα κομμάτι του χρόνου Τώρα, αν δείτε τις επιδόσεις των κρατών μελών, θα δείτε πως οι επιδόσεις κάτω από τους στόχους Βαρκελώνας δεν σημαίνουν απαραίτητα πως λείπουν οι απαραίτητες δομές. Αυτό είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε. Έχω το αγαπημένο μου παράδειγμα της περίπτωσης της Φιλανδίας. Δηλαδή η Φιλανδία δεν έχει πετύχει τους στόχους Βαρκελώνας. Είναι στο 26% αλλά στη Φιλανδία η φροντίδα των παιδιών ορίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα. Η Φιλανδία λοιπόν ακολουθεί ένα συνδυασμένο σύστημα όπου έχεις επίδομα οικιακό, δηλαδή είναι ένα επίδομα σύμφωνα με το οποίο μπορούν οι γονείς να αποφασίσουν πώς θα το χρησιμοποιήσουν όταν τελειώσει η γονική τους άδεια. Και είναι τόσο ψηλό το επίδομα αυτό, όπου ακόμα και αν υπάρχει ως κοινωνικό δικαίωμα η δομή φροντίδας παιδιών, και έχουν πρόσβαση γονείς σε τέτοιου είδους δομές, παρόλα αυτά ε, επιλέγουν κάτι διαφορετικό, άρα είναι κάτω από το 27% του στόχου. Είναι δηλαδή στο 26% όπως βλέπετε. Λοιπόν, στις βόρειες χώρες θεωρείται κοινωνικό δικαίωμα, με την εξαίρεση της Νορβηγίας, παρόλο που η Νορβηγία, η Γαλλία ε, και η Σλοβενία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πορεία επίτευξης στόχου όπου καλύπτουν τους στόχους με παρόμοιο τρόπο και έχουμε και άλλα κράτη-μέλη όπου είχαμε μια μετακίνηση προς την πλήρη απασχόληση κάτι το οποίο όμως σε μεγάλο βαθμό τροχοπέδησε λόγω της κρίσης τροχοδρόμης. Συγχωρείτε. Εκεί οι εξελίξεις είναι αρκετά περιορισμένες Έχουμε την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Τσεχία, τις χώρες του Νότου, τη Λιθουανία, όπου ακριβώς συμβαίνει αυτό που σας περιγράφω. Και φαίνεται πως ε, ένα από τα σημεία συμφόρησης για τέτοιου είδους δομές φροντίδας είναι η δυσκολία που υπάρχει του επανασχεδιασμού της φροντίδας των παιδιών ε, χρησιμοποιώντας τελείως διαφορετικές δομές λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πως μιλάμε για μια προσπάθεια να ενθαρρύνουμε τους γονείς να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Αν δει κανείς λοιπόν τη δημοσιονομική πτυχή θα δείτε πως όντως υπήρξαν κάποιες εξελίξεις, ακολουθήθηκαν διαφορετικές δε προσεγγίσεις στους ε, χώρους αυτούς ε, πολιτικής επιλογής. και όπου η προτεραιότητα δάωθηκε στην απασχόληση, όπου έγινε μια διαφορετική κατανομή του φορολογικού βάρους έτσι ώστε να επηρεάζει λιγότερο την απασχόληση, όπου η κοινωνική ασφάλιση έχει επανασχεδιαστεί έτσι ώστε να συνδυάζεται καλύτερα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, τα πράγματα άλλαξαν. Ένα από τα σλόγγαν που χρησιμοποίησαν ήταν «Η δουλειά που έχεις πρέπει να αξίζει». Και αυτό συμβαίνει και με τις δομές φροντίδες ε, που θα πρέπει με να προσφέρουν θέσεις για όλα τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να καλύπτουν και τις διαφορετικές ιδέες που έχουν στα διάφορα κράτη για το πώς πρέπει κανείς να ζει. Υπάρχει το θέμα της υπογεννητικότητας, των οικογενειακών αξιών, το ποια είναι η καλύτερη κατάσταση μέσα στην οποία ανθίζει ένα παιδί. Κάθε κράτος μέλος θέτει τους δικούς του στόχους και όλα αυτά στα πλαίσια της δικής μας πολιτικής. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις οικονομικές συνθήκες που ε, ισχύουν, ε, θα πρέπει εδώ να δούμε και το χρόνο που διαθέτουν οι γονείς για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Και πού βρίσκεται η χρυσή τομή. Νομίζω πως όλοι ακόμα την ψάχνουμε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρόλα αυτά πρέπει να σας πω πως αποφασίζουν με τελείως διαφορετικό τρόπο πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Αν δούμε λοιπόν τα συμπεράσματα, 10 κράτη-μέλη έχουν πετύχει τους στέχους του Βαρκελός με το 33% για την κατηγορία την ηλικιακή 0 με 2 έτη. Και επίσης πολλές φορές αυτές οι επίσημες δομές, επίσημες δομές με δεν είναι ε, πλήρους απασχόλησης και πολλές φορές υπάρχουν άλλου είδους δομές που αποτελούν ένα σημαντικό συμπληρωματικό στοιχείο. Τώρα, για την πολιτική στην φροντίδα των παιδιών πρέπει να επανασχεδιαστεί μεν με προτεραιότητα την απασχόληση, αλλά μέχρι κάποιο συγκεκριμένο βαθμό, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα όπως η γονιμότητα, η υπογεννητικότητα, οι οικογενειακές αξίες και οι ε, ανάγκες των παιδιών. Όλοι προσπαθούν να τονίσουν το πόσο σημαντικό είναι η απασχόληση για τους ε, γονείς. Αλλά θα πρέπει οι διάφορες δομές να είναι προσβάσιμες. Αν τάσει κανείς το μοντέλο της ε, αν εξετάσει κανείς όλες τις διαστάσεις του γενετικά ουδέτερου μοντέλου ε, απασχόλησης, θα διαπιστώσετε πως οι δομέ φροντίδα παιδιών θα αποτελούν πάντα η προτεραιότητα στη χάραξη αυτή τη πολιτικής και τώρα και στο μέλλον. Merci beaucoup pour euh, cette... Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανάλυση που κάνατε που ήταν πραγματικά πολύ πλήρη. και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε όσους το επιθυμούν στην αίθουσα για να κάνουμε μία συζήτηση. Έχουμε την κυρία Κορνέλισεν που μας έκανε κάποιες ε, παρατηρήσεις αλλά και τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι ενδεχομένως θα μας φωτίσουν για κάποιες από τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν και για τα όσα έχουν συνεισφέρει ε, η ΜΕΝ και οι ΔΕ. Λοιπόν, κυρία Κονέλη, αν έχετε το λόγο, ξέρω πως έχετε κάποιες ερωτήσεις ε, τις οποίες κρατάτε για τους εμπειρογνώμονες. Βεβαίως θα ήθελα να ακούσουμε και τους υπόλοιπους και οι οποίοι σίγουρα και αυτοί έχουν ερωτήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο στα κράτη-μέλη το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται. Και οι πολύ σημαντικές επιπτώσεις που έχουν οι επενδύσεις των κρατών μελών στο χώρο αυτό. Είμαι περίεργη, πείτε μου. Υπάρχει κάποια αντιστοιχία μεταξύ του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η φροντίδα των παιδιών από τους γονείς. Δηλαδή το κατά πόσο εάν στείλεις το παιδί σου βρεφονιπιακό είσαι κακή μητέρα ή καλή, γιατί η εμπειρία μου στις κατοχώρες ήταν πως το να χρησιμοποιείς για πάνω από 30 ώρες τέτοιου είδους δομές ε, είναι κατάπτυστο, ενώ στη Δανία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και στο Βέλγιο. Αντιστοιχεί αυτό, αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης ε, με τις προσπάθειες που κάνουν τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο προσφέρονται αυτές οι δομές είναι για να επιστρέψει ο κόσμος ε, στην εργασία ή είναι κάτι διαφορετικό. Είναι δύσκολο για τις γυναίκες. Υπάρχει μια τέτοια είδος αρνητική αντιμετώπιση αυτών των δομών από τους γονείς. Μήπως θα ήταν πιο θετική η προσέγγιση αν η κοινωνία θεωρούσε πως αποτελεί ένα κομμάτι της παιδείας και της κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. Alors, euh? Ποιος από τους εμπειρογνώμονες μας θέλει να απαντήσει. Εσείς που κοιτάξατε τις διάφορες χώρες με τις διαφορετικές επιπτώσεις, θα μπορούσατε να απαντήσετε στην κυρία Κορνέλισεν. beleid Λοιπόν, αν η πολιτική αυτή συνδυάζεται απολύτως με τις προτιμήσεις των γονέων, όχι πάντοτε, όχι απαραίτητος. Δεν πρόκειται για εύκολα συγκρίσιμα μεγέθη, όμως το παράδειγμα του τι γίνεται στην Ολλανδία, όντως υπονοεί πως η πολιτική μπορεί να προσαρμοστεί ε, στο να ακολουθεί τις προτιμήσεις και τις εργασιακές συνήθειες. Βεβαίω αυτές οι προτιμήσεις, για μια φορά ακόμα, είναι αυτές που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές επιλογές. Οπότε μιλάμε για το ποιος έκανε τα αυγό. Είναι οι προτιμήσεις των νέων γονιών που θέλουν να βρουν την ε, τέλεια ισορροπία ή έχει να κάνει με τις συνθήκες και τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί βέβαια πολλές φορές μας επιβάλλεται η πολιτική του εφικτού. Οπότε ε, νομίζω ότι πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση που επηρεάζει και επηρεάζεται ταυτόχρονα. One, thing that we did pick up, which is a bit related but a bit of an aside, is that the... Um, λοιπόν, επηρεάζονται όλα από τον τρόπο με τον οποίο και τον αριθμό με τον οποίο εκπροσωπούνται στο πολιτικό μας σύστημα οι γυναίκες. Νομίζω ότι και αυτό επηρεάζει το πώς και τι ε, συνδομές προσφέρονται. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Να μας δώσετε κάποια παραδείγματα. Ναι. Όσο πιο πολλές γυναίκες είναι βουλευτές, τόσο πιο εύκολο είναι ε, να επιχειρηματολογήσουν για αύξηση του υπερυπολογισμού για τους βρυφονιπιακούς. Νομίζω ότι από τα όσα είδα στη βιβλιογραφία μου αυτό μου έμεινε. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Alors, Madame vous vouliez intervenir. Pardon, Madame Bicérès, vous vouliez intervenir aussi. Euh, oui, je peux juste euh, vous donner quelques. Ναι, να σας δώσω κάποια στοιχεία. Στην έκθεση, στη σελίδα 12, θα δείτε ένα ακόμα γράφημα. Που δείχνει ποιο είναι το ποσοστό έγκρισης του να πηγαίνει κάθε μέρα βρεφονιπιακό ένα παιδί στην ηλικία του 0 με 2 έτη. Θα δείτε πως έχει να κάνει βεβαίως και με την ε, ύπαρξη αυτών των ε, δομών, γιατί εκεί όπου πραγματικά υπάρχει κοινωνική αποδοχή, ναι, οι γυναίκες δουλεύουν πολύ και είναι απόλυτα αποδεκτές αυτές οι δομές. Ευχαριστώ. Τέσσερις ερωτήσεις για τους εμπειρογνώμονες. Euh, και θα απαντήσει όποιο αισθάνεται πιο άνετα στι ε, ερωτήσει αυτέ. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση είχε αντίκτυπο στην ε, γυναική εργασία. Και πολύ συχνά, είτε επειδή είχαν ε, επισφαλείς συμβάσεις, είτε μερικές απασχόλησης συμβάσεις, είτε λόγω του ότι είχαν μικρούς μισθούς σε σχέση με τις δυσκολίες φύλαξη των παιδιών που αντιμετώπιζαν πολλές, βγήκαν από το χώρο απασχόλησης ε, και η κρίση δηλαδή επιτάχυνε την έξοδο των γυναικών από την εργασία. Εσείς μελετήσατε παράλληλα ε, τα στοιχεία για ζήτηση προς την ε, φροντίδα των μικρών, δηλαδή μειώθηκε και η ζήτηση φροντίδας των παιδιών επειδή οι γυναίκες σταμάτησαν να εργάζονται. Δεύτερον, ποιος από εσά έχει μελετήσει τις διαφορές ανάμεσα στην διαθεσιμότητα φροντίδας παιδιών ανάμεσα στο αγροτικό και στο αστικό περιβάλλον. Για να δούμε δηλαδή αν τελικά οι γυναίκες που εργάζονται στην Ήπεθρο έχουν τις ίδιες δυνατότητες και την ίδια πρόσβαση σε δομές φροντίδας των παιδιών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχουν στα αστικά περιβάλλοντα. Τρίτη ερώτηση. Διαστάνομαι πως η συνάδελφος Κορνέλησεν ε, ενοχοποιείται πολύ, ε, αισθάνεται πολλές ενοχές για το ότι βάζει το παιδί της στον νήπιο εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όλη μου η επαγγελματική ζωή ήταν ε, στην παιδεία και τελικά διαπιστώνουμε πως αυτή τα είδη φροντίδας είναι και μέσα κοινωνικοποίησης και δόμηση της προσωπικότητας του παιδιού. Ε, παράλληλα με αυτές τις πολιτικές που κινδύνουν τα κράτη-μέλη, ε, υπάρχει παράλληλα κάποια ανάλυση που θα μπορούσε να οδηγήσει τα κράτη αλλά και τους γονείς προς ε, την ε, επίσημη ας πούμε φροντίδα των παιδιών και να μην λέμε πια ότι πέρα από τις 30 ώρες είναι πολύ ή είναι προβολικό για ένα παιδί. Αυτή είναι η τρίτη μου ερώτηση. Και η τέταρτη μου ερώτηση, γιατί μια από εσάς έδειξε πως ε, τα ευρωπαϊκά ταμεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν ε, για την ανάπτυξη της ε, φροντίδας των παιδιών. Εσείς διαπιστώσατε από το 2008 περισσότερη ζήτηση από τα κοινωνικά ταμεία για να βοηθηθούν οι σταθμοί και κυρίως όσον αφορά ατυπικά ωράρια. Να euh, euh, σας πω για την κατάσταση της ζήτηση και ε, κατά πόσο η κρίση επηρέασε τη ζήτηση υπηρεσιών. Δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία από αυτού. διότι τα νούμερα που μετρούμε δεν είναι η ζήτηση αλλά η παρουσία στις υπηρεσίες αυτές. Τα στοιχεία είναι για το 11, σε λίγο και θα έχουμε και για το 12, οπότε δεν έχουμε μετρήσει ακριβώς τις επιπτώσεις. Για τις περιφερειακές διαφορές περίπου το ίδιο ισχύει, ότι είναι δύσκολο να έχουμε στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές ε, ανάμεσα στις χώρες, αν δούμε πούμε την Γερμανία και την Ιταλία, αλλά και για άλλες χώρες όπου μπορούμε να μιλήσω ας πω για τη Γαλλία που τη γνωρίζω καλύτερα ότι πολλές φορές και στην πόλη η ζήτηση ξεπερνά τις παροχές που υπάρχουν και όχι στην Ήπεθρο. Και όσον αφορά τα διευθυντικά ταμεία... Euh, Euh, να σας παραπέμψω σε ένα πίνακα που σας δώσαμε σε, την, αυτή την, εδώ την έκθεση που μιλάει για τα ποσά που δίνονται για τις δομές φροντίδας σε επίπεδο περιφερειακών ταμείων. Για να βελτιωθεί η ποιότητα ή η ε, παρουσία είναι δύσκολο να δούμε ακριβώς ποια ποσά επενδύθηκαν σε τέτοιου είδους μέτρα. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρο να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο υποδομών, τι έχει επενδυθεί. Merci. Est-ce qu'il y a une réponse d'un expert sur euh, la question de... Ε, και όσον αφορά την ε, προσφορά αυτών των είδων φροντίδας ε, οικοδόμηση της προσωπικότητας, την ψυχολογική οικοδόμηση του παιδιού. Ναι, βεβαίως, εσείς. Als een, als een uh, uh, econoom moet je je in dat opzicht uh, enigszins bescheiden tonen, omdat dat natuurlijk vooral ook een... Uh, een uh... Λοιπόν, ως uh, οικονομολόγος, θα πρέπει να μιλήσω πολύ προσεκτικά, γιατί εδώ μιλάτε για την ψυχολογία της ανάπτυξης. Ωστόσο, ε, διάβασα πρόσφατες μελέτες ε, στη ΣΥΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι η ποιότητα ε, των δομών υποδοχής και φροντίδας των παιδιών. Και θεωρώ πως θα ήταν πολύ εύκολο να πει κανείς πως η Βερφονιπιακή σταθμή δίνουν θετική συμβολή στην ανάπτυξη των παιδιών στις κάτω Ποτέ δεν το διαπιστώσαμε αυτό και γι' αυτό είναι και πολύ ε, ε, δύσκολο για μας γιατί θέλουμε να έχουμε τεκμηρίωση αλλά δεν την έχουμε. Μπορεί, και να μην, μπορεί να μην είναι αρνητική η επίδραση του βρεφονιχικού σταθμού, ε, αλλά μπορεί και να είναι σήμαντη, γιατί τα παιδιά πάνε λίγο. Σίγουρα όμως υπάρχουν θετικές επιπτώσεις που έχουν διαπιστωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύουμε και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Και έπειτα θα ήθελα να παρέμβω και για την πρώτη σας ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για τις επιπτώσεις της κρίσης όσον αφορά τη ζήτηση θέσεων στις βρεφορυπιακούς ε, σταθμούς. Στις κάτω χώρες διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες ε, μικρότερη, χαμηλότερης εκπαίδευσης, παιδείας, χρησιμοποιούν λιγότερο τις δομές φροντίδας των παιδιών. Και αυτό για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι ε, μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιήσουν τα άτυπα δίκτυα σε σχέση με τις πιο μορφωμένες γυναίκες γιατί αυτές συχνά χρησιμοποιούν περισσότερο την κινητικότητα μετακινούνται δηλαδή από τη μια πόλη στην άλλη σε σχέση με τους γονείς τους απομακρύνονται από τους γονείς και ένας άλλος λόγος είναι ότι οι γυναίκες χαμηλότερης μόρφωσης πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Και έπειτα οι εργασίες που οι μισθοί μάλλον που παίρνουν οι γυναίκες αυτές είναι χαμηλότεροι και άρα το κόστος ε, ε, έχει αντίκτυπο και στο, στην χρήση των δομών αυτών από τις γυναίκες. Μπορεί λοιπόν η μείωση αυτή να οφείλεται σε όλους αυτούς τους ε, ε παράγοντες ή σε συνδυασμό αυτών. Ε, Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε μία ακόμη ερώτηση και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Μπορείτε να μας πείτε ποια είστε, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Σεσίλ Νόβεν. Είμαι Γενική ε, Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών. Σας ευχαριστώ που διοργανώνετε αυτήν, αυτό το σεμινάριο. Ξέρουμε ότι ο αντίκτυπος της μη αμοιβόμενη εργασίας των γυναικών στην αμοιβόμενη εργασία των ίδιων γυναικών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γνωρίζουμε πως η στόχη της Βαρκελόνης ήταν ένα είδο. Ε, προσπάθειες όχι ιδιαίτερα επαναστατικής ε, για το Συμβούλιο να δώσει συγκεκριμένους αριθμου, αριθμητικούς στόχους, αλλά βλέπουμε πως σήμερα πως δεν τα έχουμε καταφέρει και ότι ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος, υπάρχει μια τάση σχιζοφρενική ανάμεσα στον στόχο της στρατηγικής 2020, δηλαδή να υπάρχουν 75% των γυναικών να δουλεύουν και των επενδύσεων και των πρακτικών ε, επενδύσεων ε, και του προπολογισμού ε, για τις υπηρεσίες φροντίδα των παιδιών. Όσον πέρα από τις αξίες των χωρών, αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει η επιλογή και ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρχουν και να προσφέρονται. Η ερώτησή μου λοιπόν προς τους εμπειρογνώμονες είναι η στρατηγική 2020 είναι μια γενική στρατηγική και το σημείο εισόδου για τις κοινωνικές και, και οικονομικές πολιτικές της Ένωσης σήμερα. Πώς λοιπόν να προσπαθήσουμε να επανεντάξουμε τους στόχους της Βαρκελόνης, να τους ενισχύσουμε γιατί υπάρχει και το θέμα της ε, φροντίδας των ηλικιωμένων. Μπορεί αυτό να γίνει μέσω της αναθεώρησης στρατηγικής 2020 ή μέσω της ε, ένταξης της μελέτης ε, της Κομισιόν στις συγκεκριμένες συστάσεις προς τις χώρες. έτσι ώστε να αναγκαστούν δηλαδή τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με αυτό το θέμα και να κάνουν τις προσπάθειες που πρέπει. Μάλιστα σχέση μεταξύ των, ευρωπαϊκών, των στόχων της Βαρκελόνης και των στόχων 2020. Διαστάνομαι πως απευθύνεται αυτή η ερώτηση άμεσα στην Επιτροπή, στην κυρία Μπισχέρ. Παρακαλώ κυρία Μπισχέρ. Ναι, όντως ε, προσπαθούμε να θεσπίσουμε αυτή τη σύνδεση ακόμα και αν δεν φαίνεται σαφώς ακόμη στα δικά σας μάτια. Είναι αλήθεια ωστόσο πως οι στόχοι της Βαρκελόνης ε, εντάσσονται στη στρατηγική και τα στοιχεία και η έκθεση χρησιμοποιούνται ώστε να γίνουν προτάσεις και συστάσεις μάλλον στις χώρες. 11 χώρες έλαβαν μια σύσταση που σχετίζεται με τις υπηρεσίες φροντίδας το 2013. Συνεχίζεται η ανάλυση προς αυτή την κατεύθυνση και είναι αλήθεια ότι ε, μια νέα επιβεβαίωση του στόχου σε ψηλό επίπεδο θα είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε και να ξεπεράσουμε τη σημερινή κατάσταση, γιατί είναι ένας ποσοτικός απλά στόχος και έχουν πολλά να γίνουν ακόμα στο επίπεδο ποιότητας, κόστους και πρόσβασης. Οπότε χρειαζόμαστε την στήριξη όλων σας. Ευχαριστώ. Κύριε Τεβινό, θέλετε να μιλήσετε. Ναι, αν μου το επιτρέπετε, ήθελα να σας πω κάποια στοιχεία για να απαντήσουμε τα ερωτήματα που θέσατε προηγουμένως. Λοιπόν, σχετικά με την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των παιδιών και τους τρόπους ε, φροντίδας και τις διαφορετικές δομές, να σας πω πως αν δούμε τι έχουμε στη βιβλιογραφία θα δείτε πως τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε μία διάκριση και να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε και να συγκρίνουμε την ποιότητα με την ποσότητα, με τον αριθμό των θέσεων που έχουν. Η βρεφονιπιακή. Το μεγαλύτερο τμήμα της βιβλιογραφίας τίνει να προκρίνει τις θετικές επιπτώσεις το να έχει κανείς πρόσβαση στην προσχολικής, προσχολικής, δομές προσχολικής φύλαξης ε, με ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων των παιδιών ε, που βοηθούν μετά στην σχολική, στο σχολικό βίο αλλά και στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Υπάρχει δηλαδή μια σύγκληση μεταξύ μελετών ε, που έχουν γίνει από ψυχοκοινωνιολόγους όπως επίσης και από οικονομολόγους που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι ο αριθμός ορών που παραμένει κανείς σε αυτούς τους σταθμούς. Γιατί υπάρχει αυτή η αρνητική αντιμετώπιση των γυναικών που αφήνουν τα παιδιά τους τρεις, τέσσερις μέρες την εβδομάδα. Κάποιες συγκριτικές αναλύσεις που έχουν γίνει προσπαθούν να λάβουν υπόψη αυτή την διάσταση και αυτό που φάνηκε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια αρνητική επίπτωση από τον υπερβολικό αριθμό ορών ε, που έχει περάσει κανείς στις δομές φροντίδες, αλλά αυτό γίνεται στις χώρες όπου είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα που προσφέρουν αυτές οι δομές. Για τη Δανία, για παράδειγμα, δεν παρατηρήσαμε τέτοιου είδους ε, επιπτώσεις μελέτες που έγιναν, τουλάχιστον τις συγκριτικές. Και για να κλείσουμε, η αξιολόγηση αυτού λοιπόν του αντικτύπου εξαρτάται από το τι θα συγκρίνεται μεταξύ τους. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι πως η πρόσβαση τέτοιου είδους επίσημες δομές φροντίδας, ακόμα και στις χώρες όπου είναι χαμηλής ή αβέβαιης ποιότητας, παρόλα αυτά επειδή ακριβώς επιτρέπουν στη γυναίκα να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας γρήγορα και να φέρει εισόδημα στον οικοκυριό της, ε, παρόλο που είναι κακής ποιότητας, τελικά συνεισφέρουν θετικά. Υπάρχει δηλαδή αυτό το ποιοτικό αντιστάθισμισμα. Και για τα σχόλια που ακούστηκαν για τις ανισότητες, την πρόσβαση κτλ. Για τη Γαλλία, για παράδειγμα, που γνωρίζω καλύτερα σαν περίπτωση, η Μυριέλ τα είπε. Το κριτήριο δεν θα πρέπει να είναι αν είσαι σε ε, γεωργικό ή αστικό περιβάλλον, αλλά στη σύνθεση του πληθυσμού και κυρίως σε επίπεδο συνθήκων διαβίωσης που διαφοροποιείται πάρα πολύ στη Γαλλία ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ζει κανείς και όπου υπάρχουν διαφορετικές ε, δομές φροντίδας παιδιών που ε, προσεγγίζουν κατά περίπτωση τα διάφορα ευρωπαϊκά μοντέλα. Τώρα, για την απασχόληση της γυναίκας, για την επιστροφή στη χώρα, στο χώρο εργασίας και για την ε, ανάπτυξη αυτών των δομών, βασίζομαι όχι μόνο στη γαλλική εμπειρία, αλλά και στα όσα άκουσα από τους συνομιλητές μου όταν εργαζόμουν στον ΩΣΑ για το θέμα αυτό, είναι πως στο 12 το γράφημα απεικονίζει σωστά το τι γίνεται. Οι χώρες οι οποίες προσφέρουν ένα επίπεδο πρόσβασης αρκετά υψηλό είναι οι χώρες όπου οι γυναίκες και η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας ήταν το βασικό επιχείρημα για να δημιουργηθούν αυτές οι δομές. Αυτό βοηθά και τη γεννητικότητα, για παράδειγμα. Αυτό όμως το επιχείρημα ακούστηκε περισσότερο από τις χώρες οι οποίες προσεγγίζουν περισσότερο ε, το σύστημα με τις γονικές άδειες και με τα επιδόματα τέκνων. Πάντως και στη Γαλλία αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα, ένα όριο σε αυτό το επιχείρημα για την απασχολησιμότητα των γενικών. Γιατί η συζήτηση που γίνεται στη Γαλλία που είναι για την επέκταση στο μέλλον ε, των δομών αυτών και των διαφόρων ειδών βασίζεται καταρχήν στο επιχείρημα ισότητας άντρα-γυναίκα, αλλά και στη μάχη κατά της παιδικής φτώχειας, κατά της ε, σχολικής αποτυχίας. Και κάποιες μελέτες δείχνουν πως αυτό επηρεάζει ε, και το πόσο επιτυχημένα θα μπει στο σχολικό σύστημα ένα παιδί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα επιχειρήματα είναι συμπληρωματικά και υπάρχει και μία μόχλευση όλων αυτών ε, που οδηγούν στην ισότητα των φύλων που συνδυάζεται με τα παραδοσιακά επιχειρήματα για την ανάγκη της επιστροφής των γυναικών στην εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις που βασίζεται στις ε, μελέτες που έχουν γίνει. Ας περάσουμε κατευθείαν λοιπόν στο δεύτερο σεμινάριο, στο δεύτερο εργαστήριο, όπου θα δούμε και άλλα θέματα. Τώρα, σε αυτό το δεύτερο κομμάτι, θα δούμε και τα συγκεκριμένα παραδείγματα για τις διάφορες δομές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Στις κάτω χώρες, για παράδειγμα, έχουμε και πάλι ε, την... Ε, καθηγήτρια και Πλαντέγκα και μετά θα περάσουμε να δούμε τι γίνεται στο Βέλιο, τι γίνεται στη Δανία. Η Όλγα Ραστρίγινα θα μας μιλήσει για το λετονικό μοντέλο και μετά στη Σλοβακία έχουμε την κυρία Μαγδαλένα Πίσκοβα για να κλείσουμε με τον κύριο Τευνό που θα μας μιλήσει για τη Γαλλία. Ξεκινάμε λοιπόν κάτω χώρες Γερμανία, Βέλγιο, Λετωνία, Σλοβακία, Γαλλία είναι οι χώρες που θα μας απασχολήσουν. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο χωρίς καθυστερήσεις στην καθηγήτρια Γιάννη και Πλάντεγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πάλι Ολλανδικά. Οι διαφάνειες μιλούν για δημόσιες υπηρεσίες παιδικής ε, μέρημνας στις κάτω χώρες. Και στις διαφάνειες έβαλα σε εισαγωγικά το δημόσιες και αυτό δεν το έκανα τυχαία. Το έκανα γιατί στο Ολλανδικό μοντέλο δεν υπάρχει δημόσια παιδική μέρημνα πλέον. Θα σας ε, αναφέρω σε γενικές γραμμές το μοντέλο. το 2005 τέθηκε σε ισχύ ε, νόμος για την παιδική μέρημνα. Έγιναν ε, διάφορα πειράματα ε, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και το 2005 λοιπόν τέθηκε σε ισχύ το νομοσχέδιο αυτό και παρατηρήθηκε μία μεταβολή της χρηματοδότησης. Μεταφέρθηκε από την πρόσφορα στην ζήτηση. Και αυτό, αυτή η αλλαγή έγινε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και το σκεπτικό πίσω από αυτό ήταν ότι δημιουργείται ε, μια αγορά όπου οι γονείς ζητούν υπηρεσίες παιδικής μέρημνας και όσοι προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικό τρόπο. Τώρα, η ιδιαιτερότητα των 100 χωρών είναι ότι οι γονείς είναι εκείνοι που πληρώνουν για την φροντίδα και την φύλαξη των παιδιών τους. Γι' αυτό και όσοι εργάζονται έχουν συμφέρον να είναι έτσι τα πράγματα, διότι τους δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι δομές λοιπόν παιδικής αμερίμνας είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και ε, σε γενικές γραμμές είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στους γονείς και όχι μια υπηρεσία που παρέχεται για τα παιδιά. Η αλλαγή λοιπόν στην νομοθεσία με την θέση σε ισχύ του αντίστοιχου νομοσχεδίου του 2005 είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον ε, κρατικές, ε, κρατικοί φορείς ε, παιδικής μέρημνας. Οι δομές ε, αυτές ήταν ε, είτε δωρεάν είτε επιπληρωμή. 50%, 50-50 ήταν περίπου το μερίδιο. Η ιδιαιτερότητα τώρα στο ελληνικό σύστημα και αυτό που κάνει τη διαφορά ε, όσον αφορά την κατάσταση από το 2005 και μετά είναι ότι είναι το ζήτημα της διαθεσιμότητας. Πιστεύω πως το σύστημα στις κάτω έχει λειτουργήσει αρκετά καλά, διότι οι γονείς οι οποίοι ήθελαν υπηρεσίες αφροντίδες για τα παιδιά τους ήταν μια πολύ κερδοφόρος αγορά. Είπα και νωρίτερα ότι το 2000, από το 2008 ήδη καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους της Βαρκελόνης. Και πλέον πιστεύω πως μπορούμε να μιλάμε για μια καθολική κάλυψη στις κάτω χώρες. Τα παιδιά από 2,5 ετών και πάνω βρίσκονται κυρίως σε παιδικούς σταθμούς και όχι σε διάφορες καταστάσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας, όχι σε προνήπια. Στην Σκανδιναβία από την άλλη, οι γονείς έχουν ένομο δικαίωμα στην ε, παιδική μέρημνα, αντίθετα από τις κάτω χώρες. Και αυτό ίσως το είδατε και στις ε, προηγούμενες ε, διαφάνειες. Επίσης, στις κάτω χώρες τα πάντα προσφέρονται και με δυνατότητα απασχόληση, ακριβώς όπως και οι υπηρεσίες παιδικής μέρημνας. Τώρα, η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Η ποσότητα όμως δεν έχει και τόσο καλές επιδόσεις. Η νομοθεσία αυτή του 2005 δεν ανέφερε ρητά καμία νομική ρύθμιση. Η ρύθμιση ήταν στα χέρια των ε, παρόχων. Των παρόχων και των ε, εκπρόσωπων των γονέων. Οι πάροχοι λοιπόν υπηρεσιών παιδικής εμέριμνας και οι γονείς είναι εκείνοι που παίζουν ρόλο, όμως όχι τόσο σημαντικό. Υπάρχουν λοιπόν στις κάτω χώρες ε, διάφορες ε, προδιαγραφές σχετικά με το προσωπικό, με τις ε, απολαβές, με την ποιότητα των υπηρεσιών και τις ώρες εργασίας. Τώρα, όσον αφορά την, τις πληροφορίες που έχουμε από το 2005 και μετά, έχει παρατηρηθεί μια μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών παιδικής ε, μέρημνας και αυτό εξηγείται εν μέρη από την αυξημένη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες φροντίδας ε, παιδιών η αγορά εργασίας ήταν σχετικά κλειστή μέχρι το 2005 και από το 2005 και μετά. Γι' αυτό λοιπόν οι επιδόσει είναι σχετικά χαμηλέ. Το ενδιαφέρον όμω, είναι τι έχει γίνει σχετικά με, τον λόγο απόδοση και κόστου στην αγορά εργασίας. Ε, οι αλλαγές αυτέ στόχο είχαν να επιφέρουν θετικές αλλαγές και στο θέμα του κόστους και στον ε, τομέα των υπηρεσιών υγείας. Γενικά οι αλλαγές αυτές έγιναν έτσι ώστε να βελτιωθεί η αγορά εργασίας και η παροχή των ε, υπηρεσιών. Αυτό που παρατηρήσαμε όμως ήταν μια μεγάλη αύξηση στα χρήματα που είχαν διατεθεί για τον κλάδο αυτό. Αυτό είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε το τρίτο συμβαλόμενο μέρος. Υπάρχουν δηλαδή προσφο... διάφορες προσφορές, όμως οι γονείς είναι εκείνοι που αποφασίζουν το πόσα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υπάρχουν πολύ πάροχοι υπηρεσιών ε, παιδικής εμέριμνας, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Και έχουμε παρατηρήσει επίσης μία μετάβαση από τις άτυπες στις επίσημες ε, δομές παιδικής μέρημνας. Τώρα κάτι περισσότερο τεχνικό, ε, ωστόσο εξίσου σημαντικό για να κατανοήσουμε το Ολλανδικό μοντέλο είναι το πώς οι αρχές εξετάζουν το σύστημα, το εξετάζουν βασισμένοι στην, ε, στις απολαβές ανά ώρα. Από τη στιγμή που στόχος είναι να παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες ε, ώρες υπηρεσίας ανά εβδομάδα και ανά χρόνο. Στόχος ε, είναι να υπογράφονται όσο το δυνατόν ε, μεγαλύτερες συμβάσεις. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η μετάβαση από τις άτυπες στις επίσημες δομές. Όμως αυτό επέφερε και αύξηση των ορών ε, παροχής υπηρεσιών και αυτό επιβάρυνε τον προπολογισμό. Παρατηρείται από το 2009 και μετά μια τάση περικοπών ε, στις δαπάνες μέχρι το 2012 Και επίσης έχουν περιοριστεί και έχει περιοριστεί και η άτυπη παροχή υπηρεσιών. Επίσης έχει παρατηρηθεί μια άμεση σύνθεση του πόσες ώρες έχει το παιδί σε φρεφονιπιακούς σταθμούς και τι ποιότητα υπηρεσιών έχεις. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στις 20 ε, ώρες απασχόλησης και στις 40 ώρες ε, παροχής ε, υπηρεσιών παιδικής αμέριμνας θεωρείται κάτι το πάρα πολύ αρνητικό. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν μια κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών παιδικής εμέριμνας. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν αυτή η σύνδεση ανάμεσα στον αριθμό των ωρών που εργάζεται κάποιος ανά εβδομάδα. Δηλαδή, Εάν εργάζεσαι 20 ώρες την εβδομάδα, έχεις δικαίωμα 28 ώρων παιδικής μέρημνας, επιδοτούμενης παιδικής μέρημνας. Και αυτό το ήταν κάτι που τότε δεν είχε θεωρηθεί αρκετά σημαντικό. Επιβεβαίωσε όμως ότι το μεγαλύτερο όφελος το είχε η αγορά και όχι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, τα παιδιά δηλαδή. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση των ε, τιμών και αυτό σε συνδυασμό με την ε, οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε μείωση της παροχής υπηρεσιών παιδικής μέρημνας. Και αυτό έπληξε ιδιαίτερα τις οικογένειες που έχουν χαμηλό εισόδημα, χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Τώρα βλέπουμε κάτι μη τυπικό όσον αφορά την ε, προσφορά και τη ζήτηση στο Ολλανδικό μοντέλο, όμως είναι και μια πολύ πρακτική προσέγγιση, διότι στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μοντέλο. Έχουμε εστιάσει όμως ε, σε μεγάλο όγκο προσφοράς υπηρεσιών με μειωμένη ποιότητα υπηρεσιών. Και σε σύγκριση με το βελγικό μοντέλο βλέπουμε ότι το ολλανδικό μοντέλο δεν είναι τόσο ελκυστικό. Στόχος της πολιτικής αυτής ήταν να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες για την παιδική μέρημνα και η ποιότητα όπως σας είπα είναι κάτι πάρα πολύ ε, σημαντικό και αρκετά προβληματικό στις κάτω χώρες. Και αυτό έχει άμεση σχέση με το αν οι υπηρεσίες προσφέρονται είναι, έχουν καθεστώς πλήρους ή μια απασχόλησης. Θεωρείται πως αν χρησιμοποιεί κάτι λιγότερες ώρες, η ποιότητα δεν θα είναι και τόσο καλή. Οι υπηρεσίες τέλος παιδικής ε, μερίμνας συνεχίζουν ακόμα και τώρα να θεωρούνται ως ένα, με, ως ένα από τα συστατικά στοιχεία της αγοράς εργασίας και όχι ως κάτι που σκοπός του είναι το όφελος του ίδιου του παιδιού. Σας ευχαριστώ. Merci. Pour que nous puissions garder quelques... Σας ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να έχουμε λίγα λεπτά για να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, θα ζητήσω από τους πέντε επόμενους ομιλητές να μιλήσουν μόνο για οκτώ λεπτά, παρακαλώ. Το λόγο έχει η Αλεξάνδρα Σίλε για το γερμανικό μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με χαρά μου θα σας παρουσιάσω το γερμανικό μοντέλο και θα αρχίσω αυτή εξ αρχής με δύο πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες όσο αφορά το background. Η μία έχει να κάνει με την εξέλιξη της αγοράς στη Γερμανία και η άλλη με την δημογραφική εξέλιξη στη Γερμανία. Διότι η οι υπηρεσίε παιδικής μέρημνα έχουν επικιαχυνθεί πάρα πολύ από την ε, δημογραφική αλλαγή και από την συμμετοχή των γυναικών ε, στην αγορά εργασίας. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της συμμετοχής των γυναικών ε, στην αγορά εργασίας και με καθεστω πλήρους και ιδιαίτερα με καθεστώς ήμι απασχόλησης, με αυτά στι μήνυ δουλειέ, όπω λέμε. Επίσης, η Γερμανία έχει πάρα πολύ χαμηλό αριθμό γεννήσεων, αρνητικό δημογραφικό ισοζύγιο και αυτό πλήττει ιδιαίτερα τις ε, γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση, οι οποίες συνήθω δεν κάνουν παιδιά. Τα τελευταία χρόνια η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναγνώρισε τις ε, δημογραφικές αυτές αλλαγές και τις αιτίε τους και ως αποτέλεσμα αυτών ήταν το 2007 το ένομο πλέον δικαίωμα των γονέων σε παιδικό σταθμό από τα τρία, για παιδιά ηλικίας τριών ετών και πάνω. Υπήρξε μια πολιτική λοιπόν συμφωνία υπερκομματική για αυτό και να σας πενθυμίσω εδώ ότι στη Γερμανία έχουμε ομοσπονδιακό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι παρότι η κυβέρνηση συμφώνησε για αυτό το ένομο δικαίωμα σε παιδικό σταθμό από, για παιδιά ηλικία από τριών ετών και πάνω. Η απόφαση όμως αυτή μπορεί να ε, επηρεάζει άμεσα την κατάσταση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, όμως ε, έχει ελάχιστη επιρροή σε επίπεδο κρατηδίων, τοπικό επίπεδο. Έχει παρατηρηθεί Μία αδυναμία λοιπόν από τότε που ετέθησαν αυτοί οι στόχοι τη ομοσπονδιακή κυβέρνηση να εφαρμόσει στην πράξη του στόχου η οποία η ίδια έθεσε. Τώρα, επιθυμία πέραν από την αύξηση των ε, θέσεων του παιδικού σταθμού ήταν να αυξηθεί και η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, διότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων, αλλά και υπήρξε επιθυμία να αυξηθεί το ποσοστό των γεννήσεων. Και αυτά ήταν άμεσα λοιπόν συνδεδεμένα με την απόφαση της κυβέρνηση να ε, αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα παιδικής εμέριμνας. Μετά, πολύ σημαντικό ρόλο στη Γερμανία είχε και η εκπαίδευση των παιδιών από την πρώτη παιδική ηλικία. Τώρα, Όσον αφορά τους στόχους της Βαρκελόνης, να σας πω ότι η Γερμανία εκπλήρωσε πολύ γρήγορα τους στόχους της Βαρκελόνης. Το 98% των παιδιών από ηλικίες, σε ηλικίες τριών ετών και πάνω βρίσκονται ήδη σε κάποιο παιδικό σταθμό. Ωστόσο, Όπως είπαν και οι προηγούμενες ομιλήτριες, οι θέσεις αυτές στους παιδικούς σταθμούς είναι θέσεις ήμι απασχόλησης. Η, η συμμετοχή σε επίσημους ε, παιδικούς σταθμούς είναι στο 29,3%. Επίσης, Η Γερμανία δεν είναι μόνο μια ομοσπονδιακή δημοκρατία, αλλά αποτελείται και από, την, από δύο κομμάτια, από την Δυτική και την πρώην Ανατολική Γερμανία. Και εκεί παρατηρούνται μεγάλες διαφορές, λοιπόν. Στην Δυτική Γερμανία το 2011 20% των παιδιών ηλικία κάτω των 3 ετών βρίσκονταν σε, κάποια, σε κάποιο παιδικό βρεφονιπιακό σταθμό. Στην Ανατολική Γερμανία το ποσοστό όμως αυτό ήταν κατά πολύ μικρότερο. Και εμείς αυτό το έχουμε θεωρήσει ως ένα αποτέλεσμα των πολιτισμικών διαφορών στην Ανατολική και στην Δυτική η Γερμανία. Είναι ακόμα ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα το να εργάζεται μία μητέρα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και ταυτόχρονα να έχει τα παιδιά της όλη τη μέρα σε έναν βρεφονιπιακό σταθμό. Αυτό η Ανατολική Γερμανία όμως έχει ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα ίσως πιο ανεπτυγμένο όσον αφορά την ε, παιδική μέρημνα και τη συσχέτισή της με την απασχόληση. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι διαφορές και όταν μιλάμε για τη Γερμανία πρέπει να δούμε όλες τις ε, συνιστώσεις της τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα, τις γεωγραφικές διαφορές, το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται. Επίσης αναφέρθηκε και πιο πριν ότι υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές από κρατήδιο σε κρατήδιο. Υπάρχουν, για παράδειγμα, πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη Βαβαρία, που είναι ένα πολύ μεγάλο κρατήδιο, και σε πόλεις κρατήδια, όπως το Αμβούργο και το Βερολίνο ή η Βρέμη. Στη Γερμανία λοιπόν υπάρχει μια αρκετά τερογενής ε, προσφορά υπηρεσιών παιδικής εμέριμνας. Καταρχάς υπάρχουν διαφορές από κρατήδιο σε κρατήδιο. Αυτό οφείλεται στην νομοθεσία και στο πώς αυτή εφαρμόστηκε και στο πόσο γρήγορα εφαρμόστηκε, στα κονδύλια που διατίθενται και στο χαρακτήρα των υπηρεσιών και των βρεφονιπιακών σταθμών. Το 1 τρίτο μόνο είναι κρατική φορείς, τα δύο τρίτα όχι. Και αυτό το ονομάζουμε εμείς σε πλουραλισμό της παροχής. Σε πολλοί βρεφονιπιακοί σταθμοί συντηρούνται από την Εκκλησία, από, δια, από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή από εθελοντικές οργανώσεις. Επίσης, πολλές δομές στηρίζονται όχι από το ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά από το τοπικό επίπεδο. Και οι γονείς συνεισφέρουν, οι γονείς πληρώνουν για, την, για μια θέση στον Ευρωφωνηπιακό Σταθμό. Υπάρχουν λοιπόν ε, εδώ διακυμάνσεις στις τιμές, οι οποίες έχουν να κάνουν και με το εισόδημα των γονέων, αλλά και με το αν ένας βρεφονιπιακός σταθμός είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, ή και το τι προσφέρει, αν είναι ένας απλός βρεφονιπιακός σταθμός ή αν προσφέρει και μαθήματα μουσικής, για παράδειγμα. Επίσης υπάρχουν διάφορα στάνταρτ όσον, αφορά ε, όσον αφορά την ποιότητα την ποιότητα ε, και τις ε, δεξιότητες του προσωπικού που απασχολείται σε αυτούς τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Εάν αυτοί οι υπάλληλοι έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στις μεγάλες διαφορές ε, που παρατηρούνται στη Γερμανία. Επίσης, ένας από τους άλλους παράγοντες με τους οποίους υπολογίζουμε την ποιότητα είναι το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι γονείς από τις υπηρεσίες ε, παιδικής μερίμνας που τους ε, παρέχονται. Έχουν γίνει πάρα πολλές, πάρα πολλές έρευνες αυτό. με τις οποίες προσπαθούμε να δούμε τη σχέση με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. Τώρα, οι δομές κρατικές σημεί είναι μία από τις ε, συνιστώσεις. Ενδιαφέρον όμως επίσης είναι ότι στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχουν ε, εισαχθεί πολλά μέτρα τα οποία έχουν επηρεάσει την ε, συσχέτιση οικογένειας-εργασίας. Καταρχάς τα διάφορα ε, επιδόματα και διάφορες ε, άδειες. Η γονική άδεια, για παράδειγμα, είναι ένα μέτρο που έχει εισαχθεί. Τα επιδόματα τέκνων επίσης, τα οποία εξαρτώνται από το εισόδημα της κάθε οικογένειας. Επίσης το επίδομα για κατοίκον φύλαξη τέκνου, το οποίο δεν αντικαθιστά βέβαια τον, ε, έναν μισθό. Είναι όμως ένα πρόσθετο μέτρο που έχει στόχο να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Προσπαθούμε σε αυτό το θέμα να ακολουθήσουμε κάπως το σκανδιναβικό μοντέλο, το σουηδικό μοντέλο. Με το να δίνουμε το δικαίωμα και στους δύο γονείς να παίρνουν γονική άδεια. 12 μήνες για τον ε, ένα γονέα και δύο μήνες παραπάνω για τον δεύτερο. Επίσης, ένα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα στη Γερμανία είναι ε, το ένομο δικαίωμα λοιπόν των ε, γονέων για μια θέση σε παιδικό σταθμό από το 2007. Αυτό ήταν μια συμφωνία, όπως σας είπα, υπερκομματική το θέμα όμως αυτό παραμένει αμφιλεγόμενο και παραμένει αμφιλεγόμενο διότι μαζί με αυτό το μέτρο εισήχθηκε ένα νέο επίδομα, το επίδομα κατοίκων φύλαξης τέκνου, το οποίο μάλιστα είναι από τον Αύγουστο του 2013 νόμος το επίδομα λοιπόν αυτό είναι ύψους 100 ευρώ και το λαμβάνει ένας εγωνέας εάν έχει παιδί κάτω από τριών ετών, το οποίο δεν το στέλνει σε βρεφονοπιακό σταθμό, αλλά το φροντίζει στο σπίτι του. Και είναι ένα πραγματικά αμφιλεκόμενο θέμα για το, όσον αφορά το πόσο ωφέλιμο είναι, το πόσο βοηθά τους γονείς ή το παιδί. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα τα επιδόματα αυτά με την οικογενειακή πολιτική που προσπαθούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον ε, Γιάνν Πίτερς να μας εξηγήσει την περίπτωση του Βελγίου. Είμαστε κι εμείς ε, ομοσπονδία, το οποίο σημαίνει πως και η προσχολική αγωγή αλλά και η βρεφονιπιακή ηλικία ε, αποφασίζονται από τις ε, δύο διαφορετικές κοινότητες, αλλά νομίζω ότι ακολουθούν παρόμοιες πορείες. Παρόλο που είχαμε αρκετές συστάσεις από διεθνείς οργανώσεις, το Βέλιο αποφάσισε να μην εντάξει τις βρυφονιπιακές δομές στις ε, σχολικές δομές. Είμαστε ένα από τα δύο κράτη που έχει πετύχει το 99% ε, των παιδιών μεταξύ 2,5 και 6 ετών να έχουν θέση σε τέτοιου είδους δομές και για το 0 με 3 το 38%. Και Αντίθετα με τη συζήτηση που έχει γίνει σήμερα, παρόλη την οικονομική κρίση, δεν είχαμε μείωση των αριθμών που προσφέρονται, αντίθετα, των αριθμών θέσεων που προσφέρονται, αντίθετα έχουν αυξηθεί αυτές. Έχουμε φτάσει δηλαδή σήμερα στο 38% από το 32% στο 2008. Το 2010-2011 είδαμε μια αύξηση στον αριθμό θέσεων ε, της τάξης του 3 περίπου σε κάθε ε, μία από τις δύο κοινότητες. Η φλαμανδική κοινότητα έχει φιλόδοξους στόχους, θέλει 50% των παιδιών σε αυτή την ηλικία να έχουν θέσει σε ευρωφωνηπιακό σταθμό και για τις Βρυξέλλες ε, προσπαθούν να δημιουργήσουν 60.000 επιπλέον θέσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι πως η ανεργία στη γυναίκα ε, στο Βέλγιο από την απαρχή της κρίσης μειώθηκε. Είναι 7,4% σήμερα, ήταν 8,5% το 2008. Και παρόλα αυτά έχει φτάσει το 7, κάτι από το 6,1% που ήταν στους άντρες. Άρα λοιπόν αυτή η προσφορά τέτοιων θέσεων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς έχει ωφελήσει τη γυναικεία απασχολησιμότητα. Πάντοτε είχε και παιδαγωγικό ρόλο αυτή η αγωγή. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι πως οι πολιτικοί στις τρεις ε, κοινότητες ουσιαστικά ανταποκρίνεται ε, σε όλους τους στόχους ε, αυτής της αγωγής. Δηλαδή οικονομικό, η γυναίκα πίσω στη δουλειά, ε, διδακτικό, τα παιδιά να μαθαίνουν, αλλά και κοινωνικό, δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες και ίσες ευκαιρίες για όσους μεγαλώνουν σε περιοχές με μειονεκτήματα. Δεν θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που λένε πως δεν υπάρχουν εμπειρικές ή επιστημονικές μελέτες που να αποδεικνύουν πως δεν είναι καλές αυτές οι δομές για τα παιδιά. Εγώ πρέπει να σας πω πως για την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχω κάνει πάρα πολλές μελέτες και πρέπει να σας πω πως είναι πολλά τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν πόσο θετικό είναι ο αντίκτυπος αυτών των δομών στα παιδιά, κυρίως που μεγαλώνουν σε οικογένειες που μειονεκτούν. Δηλαδή προσφέρουν ευκαιρίες στα παιδιά αυτά. Τώρα, αν εξετάσει κανεί τι τρεις κοινότητες, θα δει πω η Φλάνδρα πάνω απ' όλα, η φλαμανδική κοινότητα, έχει εξετάσει περισσότερο την κοινωνική διάσταση. Δηλαδή, δημιούργησαν τέτοιου είδου δομέ έτσι ώστε να υπάρχει ε, απόλυτη ε, πρόσβαση και έχουν ε, ε και κονδύλια έτσι ώστε να έχουν δυνατότητα πρόσβασης και οι πιο φτωχοί Υπάρχει μια στοχευμένη προσέγγιση που ακολουθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ξέρετε πω στην επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρεται ω πολιτική που θα έπρεπε να επιτρέπει πρόσβαση σε όλου και όχι με ισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, για όλου, Και όταν λέμε για όλου εννοούμε και αυτού από ε, που μειονεκτούν. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι οι ίσε ευκαιρίες στην παιδεία. Δηλαδή η χρηματοδότηση των νηπιαγωγείων και των δημοτικών που έγινε σύμφωνα και με τους στόχους που είχαν τεθεί πέτυχε. Όσα πιο πολλά παιδιά βρίσκονται σε ένα σχολείο από υπόβαθρα που μειονεκτούν, τόσο πιο πολλά χρήματα ελάμβανε το σχολείο αυτό από τον κεντρικό προϋπολογισμό και όλες οι χώρες, με συγχωρείτε και όλες οι θέσεις ε, στους βρεφονιπιακούς σταθμούς είχαν κρατηθεί για όσους ε, είναι πιο φτωχοί. Αντίθετα, στην Βαλονία το είδαν πιο εκπαιδευτικά. Και βλέπετε ότι το, στην ηλικία 0 με 3 έχουν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο που συνδυάζει και τη συμμετοχή της οικογένειας με βασικούς παιδαγωγικούς στόχους ε, για την περιοχή των Βρυξελών και τη Βαλονία. Και γίνεται μια επιθεώρηση των στόχων αυτών με πολύ στενό τρόπο. Πρόκειται παλιά για μια απλή παρακολούθηση. Σήμερα μιλάμε για την παιδαγωγική εξέλιξη και την παιδαγωγική προγύμναση αυτών των νηπίων Η ποιότητα λοιπόν αυτή τη παρεχόμενη φροντίδα είναι αυτό που του απασχολεί. Στο Βέλγιο οι γυναίκε έχουν 15 εβδομάδε γονική άδεια και από το 2003 έχουν και οι οι πατεράδες 10 μέρες και κάθε ένας μπορεί να πάρει και κάθε χρόνο 3 μήνες μέχρι το, ε, τα έκτα γενέθλια του παιδιού. Τώρα, τα επιδόματα είναι ακόμα κεντρικά, αλλά στο μέλλον θα τα αναλάβουν οι ε, δύο κοινότητες, οι τρεις κοινότητες. Είναι αρκετά γενναιόδρα τα επιδόματα αυτά, δηλαδή αν έχεις τρία παιδιά, ε, λαμβάνεις 500 ευρώ το μήνα. Και διάφορες έρευνες εξήγησαν πως γι' αυτό ακριβώς έχουμε πολύ λίγα παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας στη Βέλγιο σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως θα πρέπει να, ε, υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια και να πληρώνουν ε, το όριο είναι τα 32 ευρώ την ημέρα και βεβαίως μπορούν και τα ε, έξοδα αυτά μέχρι τα 11 ευρώ την ημέρα να τα δηλώνουν ως έξοδα στη φορολογική τους δήλωση. Το βολγικό μοντέλο λοιπόν βασίζεται στην προσβασιμότητα και την προσπελασιμότητα ε, σε αυτές τις θέσεις και στα γενναιόδερα επιδόματα. Τώρα, ε, γεννητικότητα. Είμαστε πολύ πάνω από το Ευρωπαϊκό Μέσο του 1,4. Εμείς είμαστε πάνω από το 1,9 παιδιά ανά οικογένεια. Και παρόλη την κρίση και οι τρεις κινούντες επενδύουν στην αύξηση των ε, θέσεων. Έχουμε μια ποιοτική παράδοση και παρακολουθούμε την διάσταση ποιότητας και για την προσχολική ηλικία και για την βρεφονιπιακή. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό ξεκίνησε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις Βρυξέλλες θα εγκριθεί ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα έτσι ώστε να βαθμολογούν την ποιότητα τα παιδιά και οι γονείς. Και σε όλες τις κοινότητες είδαμε να γίνονται πολλές επενδύσεις στην ποιότητα της ε, φροντίδας των παιδιών. Και στη Φλάνδρα υιοθετήθηκε ένας νέος νόμος που εξετάζει και την επαγγελματική πορεία όσων ε, ε, εργάζονται σε, αυτούς, αυτές τις δομές. Να σας πω τέλος πως οποιοδήποτε εργάζεται στην ε, βρεφονιπιακή ε, και στην νηπιακή φροντίδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πτυχίο νότο του Ιδρύματος. Βέβαια δεν είναι όλα ρόδινα. Μια μελέτη της UNESCO έδειξε πως η χώρα η οποία ενσωματώνει ε, τα νηπιαγωγεία στο σχολικό σύστημα δίνει ένα πλεονέκτημα. Και βεβαίως οι εργασιακές συνθήκες βελτιώνονται και βελτιώνονται και τα επαγγελματικά προσόντα των όσων εργάζονται στους σταθμούς αυτούς, κάτι το οποίο τους κάνει πιο ποιοτικού τελικά. Αν δει κανείς δηλαδή τι συμβαίνει όταν τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στο σχολικό σύστημα, θα δείτε πως και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 δίνεται μια παρότρινση να γίνει αυτό. Πρέπει να σας πω πως στην ε, φλαμανδική κοινότητα είναι πολύ ανειδίκευτη, για να τους πούμε έτσι, που εργάζονται σε αυτούς τους βρεφονιπιακούς ε, σταθμούς και είπαν πως μέχρι το 2024 θα πρέπει όλοι να έχουν ειδική εκπαίδευση. Για την προσχολική εκπαίδευση είδαμε πως τα πιο μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα και Το πρόβλημα είναι ότι είναι με πολλά τα παιδιά συντάξει, 20 με 25 παιδιά ε, αναδάσκαλο Κάτι το οποίο έχει πολύ ε, αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξή τους. Και βεβαίως έχουμε πολλές αποκλήσεις. Στις Βρυξέλλες, αν ρίξετε μια ματιά, θα δείτε, θα δείτε οι γονείς πολλές φορές ως ε, σύλλογοι γονέων κάνουν και αυτοί παράλληλα προσπάθειες. Ε, ε, και τώρα θα ακούσουμε την κυρία Όλγα Ραστρίτζινα που, για την Λετωνία. 8 λεπτά έχετε και μετά Σλοβακία και Γαλλία. 3-8-24 κάμε. κάνει. έχουμε αργήσει. Παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στο χρόνο που σας έδωσα. Good afternoon. Uh, I'm going to present uh, the Latvian model um, of care provision. Να σας, θα σας μιλήσω για την μέρημνα για τα παιδιά, όπως προβλέπετε στην Λετωνία, που χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό απασχόλησης των γυναικών. Από τη μια πλευρά αυτή είναι μια θετική, ένα θετικό κληροδότημα της Σοβιετικής περίοδου, που οι γυναίκες δούλευαν το ίδιο με τους άντρες, και από την άλλη ε, το πρότυπο αυτό παραμένει ανάγκη, διότι... Ε, η, ε, ε, χρειάζεται, τα, τα ημερομήνες είναι χαμηλά και χρειάζεται να εργάζονται ε, και οι γυναίκες. Ε, οι μερικέ απασχόλησει θέσει δεν υπάρχουν πολύ και δεν είναι και συμβατέ πολύ με ψηλέ αμοιβέ. Επίση δεν είναι διαδεδομένε οι ευέλικτε μορφέ εργασία. Αυτό καθιστά δύσκολο το συνδυασμό με την οικογενειακή ζωή, ιδιαίτερα για τους ε, γονείς μικρών παιδιών. Οι δημογραφικές εξελίξεις επίσης στη Λετωνία δεν είναι πολύ θετικέ. Έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητα στην Ένωση. Επίσης ε, η Λετωνία χτυπήθηκε από διάφορα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα από την ε, εξαρτησία της και μετά. Καταρχήν στη δεκαετία του 90 μετά την είσοδο στην Ένωση και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Ε, σύμφωνα με τις τελευταίες δημογραφικές εξελίξεις, ακόμα και με το πιο θετικό σενάριο, το νούμερο των παιδιών που γεννιέται κάθε χρόνο θα μειώνεται, θα βαίνει μειούμενο στις επόμενες δεκαετίες. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια, η φροντίδα των παιδιών για να μπορούν οι γονείς να είναι πιο άνετοι, αλλά και να μπορέσει να προωθηθεί η γονιμότητα και η γεννητικότητα. It's, um, Latvia's development has been quite limited, especially for children below three years old. In 2011... Λοιπόν, το 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαμε, μόνο το, 15, το 50%, ε, συγγνώμη, το 15% των παιδιών ε, ε, ε, καλύπτονταν από τις δομές που είχαμε και εδώ με τις στάσεις από το 2005 η πρόοδος ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Performance with respect to the second target Uh, was more positive in 2000... Τώρα, δεύτερο στόχο στόχος της πιο θετικά τα πράγματα. Το 2007 το 73% ηλικίες 0 μέχρι 3 ετών καλύπτονταν από τη φροντίδα των παιδιών, τι δομέ, αλλά και πάλι είμαστε πιο κάτω από το στόχο και αν δείτε το γράφημα, τα περισσότερα παιδιά ε, καλύπτονται full time, πράγμα το οποίο είναι συμβατό με τις ώρες απασχόλησης των γονέων. Πώς οργανώνεται τώρα η φροντίδα των παιδιών στη Λετωνία. Ιστορικώς η φροντίδα των παιδιών ενσωματώνεται στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρώτη νομοθεσία περί ε, παιδείας συμπεριλάμβανε την ε, βρεφιονιβιακή φροντίδα τα περισσότερα σχολεία έχουν και βρεφονιβιακούς σταθμούς. Για τα παιδιά μέχρι 4 ετών είναι θελοντική φίτηση, ενώ από τα 4 και μετά είναι υποχρεωτική. Στα 7 αρχίζει η βασική εκπαίδευση, το δημοτικό. Αυτή τη στιγμή οι, οι ιδιώτες ε, πάροχοι φροντίδας των παιδιών είναι σπάνιοι, ιδιαίτερα αυτό που δεν, που δεν έχουν κάποια εκπαιδευτική πτυχή, όπως ας πούμε Βρεφονιμπιακή που είναι διαθέσιμη μόνο για το πρωί ας πούμε δεν είναι συμβατή με το πλήρες ωράριο των γονέων. Το ιδιωτικό τομέα ε, συμβαδίζει με τον δημόσιο στις παροχές του. Οργανώνεται λοιπόν η φροντίδα των παιδιών από την τοπική κυβέρνηση. Για τα παιδιά μέχρι τα τέσσερα οι τοπικέ κυβερνήσει είναι υποχρεωμένε να εξασφαλίζουν την ίση πρόσβαση. Ωστόσο αυτό ο στόχο δεν επιτυγχάνεται λόγω των περιορισμένων ε, δημοσιονομικών πόρων σε κάποιου Δήμου. Για τα παιδιά από τα 4 μέχρι τα 6 οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να εγγυώνται δωρεάν θέσει στο νηπιαγωγείο. Οπότε σε αυτή την ε, ηλικιακή ομάδα δίνεται προτεραιότητα αν υπάρχουν ε, λιγοστέ θέσει. Οπότε πρέπει να είναι καθολικό το σύστημα στη Λετωνία ε, να καλύπτουν όλα τα παιδιά, αλλά λόγω των οικονομικών δυσκολιών δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Ωστόσο, υπάρχει παροχή περιδιδικής μέρημνας κατοίκων με σχεδόν μηδενικό κόστος. Τώρα, από το 2013 συγχρηματοδοτείται η φροντίδα των παιδιών για τα παιδιά από 1,5 μέχρι 4 ετών, η ιδιωτική μάλιστα κάλυψη και υπάρχουν ε, και κάποιες ε, ε, πιο χαλαρές ρυθμίσεις για την ιδιωτική παροχή μέρημνας για τα παιδιά. Τώρα θα πρέπει να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι τάσεις, μάλλον οι προβλέψεις και αν είναι θετικός αντίκτυπος για την μέρη με το παιδιά. Τώρα, τάσεις και κάλυψη. Όπως ξέρετε η Λετωνία χτυπήθηκε πολύ ε, σοβαρά από την οικονομική κρίση. Το ΑΕΠ έπεσε κατά πάνω από 25%. Ωστόσο δεν είδαμε μεγάλη επιρροή της κρίσης στην παροχή της φροντίδας των παιδιών και γι' αυτό γιατί ταυτόχρονα οι υποδομές των, νηπίων, των νηπιαγωγείων είχε ήδη βελτιωθεί μέσω της στήριξης του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου. Ωστόσο, δεν ανταποκρινόμαστε σε όλη τη ζήτηση. Το 2011, 67,8% των παιδιών καλύφθηκαν για την ηλικία 1,5 μέχρι 6 έτη και το 8,8% ήταν στη λίστα αναμονής και αυτά με βάση τις εθνικές μας, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μας. Τώρα, να αναφέρω ότι διαχρονικά αυξήθηκε η κάλυψη ε, της μέρημνας των παιδιών, αλλά αυτό οφείλεται βασικά στην αλλαγή της δημογραφικής δομής του πληθυσμού, δηλαδή μείωση της γεννητικότητας. Τώρα, συμπληρωματικά μέσα, μέτρα, ε, είναι βασικά τα επιδόματα αναπαιδεί. Έπειτα έχουμε τα 70 με 80% του μέσου, ε, της μέσης αμοιβή είναι τα επιδόματα μητρότητας ή πατρότητας, ε, τα γονικά επιδόματα. Αν κάποιο γονιό δεν είναι πλέξιμο για τα επιδόματα αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα επίδομα παιδί που είναι συγκεκριμένο ποσό αναμήνα. Όταν το παιδί φτάσει το ένα έτος ή το 1,5 έτος, τότε η οικονομική στήριξη από την κυβέρνηση μειούται πολύ γρήγορα. Και σε αυτή τη φάση συνήθως οι γονείς πρέπει να επιστρέψουν και στην ε, δουλειά τους. Το 2014 αναμένονται διάφορες αλλαγές. Καταρχήν το ποσοστό κατάργησης των γονικών επιδομάτων θα μειωθεί και θα μειωθούν δηλαδή έτσι τα κίνητρα για να επιστρέφουν οι γονείς στην δουλειά τους. Και επίσης θα αυξηθούν τα μίνιμουμ ποσά για τα παιδικά επιδόματα για τα παιδιά μέχρι 5 ετών. Να τονίσουμε πως ε, η εργασιακή ζωή ε, και η οικογενειακή ζωή και η ισορροπία μεταξύ τους πρέπει να βελτιωθούν. Ε, χρειάζονται λύσεις ε, πηγόντως και βραχυπρόθεσμα για τα παιδιά μέχρι 4 ετών, γιατί σύμφωνα με τις δημογραφικές τάσεις ο αριθμός των παιδιών θα μειωθεί γρήγορα και μέχρι το 2020 και μάλιστα θα φτάσει στον ίδιο νούμερο όπως ο αριθμός που τα παιδιά των παιδιών που τώρα καλύπτονται από το σύστημα. Κάποια βήματα έγιναν το 2013 για να βρεθούν αυτές οι λύσεις. Όμως αυτές οι πολιτικές χρειάζεται να αξιολογηθούν πολύ προσεκτικά και θα ήθελα επίσης να τονίσω πως δεν πρόκειται μόνο την εξασφάλιση της ίσης πρόσβασης, της πρόσβασης αλλά και την ίση ποιότητα που γενικά παραμελείται στη δημόσια συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ρωτήσουμε τους Δερμηνείς αν μπορούν να μας δώσουν πέντε λεπτά. Και θα περάσουμε άμεσα στην εμπειρία της Σλοβακίας με την ε, καθηγήτρια Πίσκοβα από την Πρατισλάβα. Παρακαλώ Πολύ έξι λεπτά μόνο να μιλήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολυτέλεια αυτή που μου δίνεται να μπορέσω να μιλήσω σλοβακικά. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή την ευκαιρία που έχω για διερμηνία. Δεν θα σας κουράσω με τις διαφάνειες και θα είμαι σύντομη. Η Σλοβακία λοιπόν ήταν μία από τις χώρες που δεν ε, κατάφερε να φτάσει στους στόχους της Βαρκελόνης. Ούτε για τα παιδιά από 3 έως 6 ετών, ούτε για τα παιδιά μέχρι 3 ετών. Και ποιος είναι ο λόγος για αυτό, ποιο είναι το πλαίσιο δηλαδή το οποίο οφείλεται. Όσον αφορά τον, ε, το ποσοστό απασχόλησης στη Σλοβακία, να σας πω ότι για τις γυναίκες το ποσοστό, απασχόληση είναι κάτω του μέσου όρου και οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι εάν το ποσοστό απασχόλησης ε, των γυναικών στη Σλοβακία φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα ανέβει το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται κατά 6% τώρα, όπως και στην Λετωνία, έτσι και στη Σλοβακία, περισσότερες γυναίκε έχουν καθεστώ πλήρους απασχόλησης όταν εργάζονται. Και όσον αφορά την ίμια απασχόληση δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί οι παράγοντες έχουν επηρεάσει λοιπόν την κατάσταση ε, με τις υπηρεσίες παιδικής εμέριμνας στη Σλοβακία, ιδιαίτερα για τα παιδιά μέχρι τριών ετών. Δεν έχουμε καθόλου θετικά αποτελέσματα λοιπόν για την ηλικιακή αυτή ομάδα. Και να σας πω ότι για την κοινωνία της Σλοβακίας μια καλή μητέρα είναι εκείνη που μένει στο σπίτι με το παιδί της τουλάχιστον μέχρι το παιδί να φτάσει τα τρία χρόνια. Χρησιμοποιεί δηλαδή όλες τις δυνατότητες γονικής άδειας, άδειας μητρότητας και η άδεια αυτή πολλές φορές φτάνει μέχρι το, τα έξι έτη του παιδιού. Αυτή είναι μια καλή μητέρα στη Σλοβακία. Η μητέρα λοιπόν πηγαίνει μετά τα έξι χρόνια του παιδιού της, ε, επιστρέφει στην αγορά εργασίας και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο μια γυναίκα να επιστρέψει στην αγορά εργασίας. Τώρα όσον αφορά τις ε, δομές που υπάρχουν, να σας πω ότι υπάρχουν ελάχιστα κέντρα ε, παιδικής εμέριμνας για παιδιά από ενός μέχρι τριών ετών. Δυστυχώς και δυστυχώ τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε δεν είναι και απόλυτα ε, αξιόπιστα με την έννοια ότι συλλέχθηκαν το 2010 και το δείγμα που ε, χρησιμοποίησαμε ήταν αρκετά μικρό, όχι επομένως αντιπροσωπευτικό. Και είναι επίσης, ε, ένα, και επίσης δεδομένα τα οποία είναι δύσκολο να επαληθευτούν. διότι οι εγκαταστάσεις ε, βρεφονιπιακών σταθμών για τα παιδιά μέχρι τριών ετών δεν ε, υπάγονται σε κάποιο επίσημο φορέα, δεν υπάγονται στο Υπουργείο ε, Υγείας πλέον όπως το παρελθόν. Η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας και, ε, Εργασίας συγγνώμη, και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα κενό και οι βρεφονιπιακοί αυτοί οι σταθμοί συνέχισαν να λειτουργούν εξαιτία της καλής εθέλησης των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούσαν. Βέβαια υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι προσπάθησαν να βελτιώσουν την κατάσταση όσον αφορά την ε, προσφορά να σας πω ότι πέραν από τις προδιαγραφές σχετικά με την υγιεινή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τους βραφονιπιακούς σταθμούς. Έτσι λοιπόν έχει κατάσταση για τα παιδιά μέχρι τριών ετών τώρα, για τα παιδιά από τριών έως έξι ετών. Βλέπετε στον ε, πίνακα την αλλαγή. Το 2003 η θάνατη ήταν για πρώτη φορά περισσότεροι από τις γεννήσεις. Υπάρχει λοιπόν υπογεννητικότητα. Ε, τώρα παρατηρείται μια πολύ αργή ανάκαμψη των γεννήσεων. Τα τελευταία δύο περίπου χρόνια Επίσης παρατηρείται και μία αύξηση του ποσοστού των παιδιών που πηγαίνουν σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Επίσης να σας πω ότι στη Σκλοβακία υπάρχουν πάρα πολλές ε, διαφορές ε, από μέρος σε μέρος. Τα σοβαρότερα προβλήματα τα αντιμετωπίζει η Μπρατισλάβα, η περιοχή της πρωτεύουσα, η οποία έχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας και το ψηλότερο ποσοστό ζήτησης. Το, χαμηλότερο, το μικρότερο πρόβλημα το έχουν οι περιφέρειες. Υπάρχει λοιπόν ένας αρνητικός συσχετισμός ανάμεσα στο ποσοστό ανεργίας και στην ζήτηση για βρεφονιπιακούς σταθμούς και για θέσεις αυτούς. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς έχει κατάσταση στις 8 διαφορετικές περιφέρειες της Σλοβακίας. Βλέπετε τι γίνεται στην Πρατισλάβα. Ε, ο αριθμός ε, των απορρι... απορριφθήσεων αιτήσεων ήταν πάρα πολύ μεγάλος σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της Σλοβακίας, όπου υπάρχει με μια έλλειψη θέσεων, αλλά δεν είναι τόσο έντονη όσο στην Πρατισλάβα, όπου απορρίπτονται αιτήσει για εισαγωγή και εγγραφή του παιδιού σε παιδικό σταθμό. Στο ανατολικό μέρος της Σλοβακίας ε, υπάρχει η μεγαλύτερη ανεργία, πάνω από 30% σε ορισμένες περιπτώσεις και εκεί παρατηρούμε ότι οι αιτήσει για ένταξη σε βρεφονιπιακό σταθμό που απορρίφθηκαν δεν είναι τόσο πολλέ. Στην Πρατισλάβα λοιπόν υπάρχει το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που είναι καλό, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό αιτήσεων που έχουν απορριφθεί, το οποίο δεν είναι καλό. Όσον αφορά τους στόχους της Βαρκελόνης τώρα, για τα παιδιά μέχρι τριών ετών, και αυτό που θα πω δεν είναι δική μου άποψη, έχω μιλήσει με τους αρμόδιους του ε, Υπουργείου. Να σας πω ότι δεν είναι ρεαλιστική επιτεύξη των στόχων, αυτών για εμάς μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν κάποιες ε, υποδομές και υποστηρικτικές δομές που μόλις τώρα έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έπειτα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συνεισφέρουν σε αυτό, οι μεγάλες διαφορές όπως είπα ανάμεσα στις περιφέρειες της ε, Σλοβακίας και οι δημογραφικές εξελίξεις, οι δημογραφικές αλλαγές οι οποίες παρουσίασαν ιδιαίτερη αστάθεια τα τελευταία χρόνια. Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια είχαμε μια θετική εξέλιξη, όμως ε, αυτό προβλέπεται να συνεχιστεί μόνο μέχρι το 2016 έως 2017. Αυτό λοιπόν εξαρτάται άμεσα με το πώς κονδύλια είναι διατεθειμένο το κράτος να διαθέσει στον τομέα της παιδικής εμέριμνας. Τέλος, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με, τη, με τους πληθυσμούς των Ρωμά στη Σλοβακία. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά το ποσοστό των παιδιών Ρωμά που βρίσκονται σε ευρεφονιπιακούς σταθμούς, όμως ε, όλες τους αυτές δείχνουν ότι μόνο το 25% των παιδιών Ρωμά βρίσκονται σε κάποιον ε, βρεφονιπιακό σταθμό. αυτό ε, λοιπόν είναι ένας ακόμα παράγοντας ε, που επιδεινώνει την ε, στατιστική μελέτη στη Σλοβακία. Σας ευχαριστώ λοιπόν για το χρόνο που μου διαθέσατε. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε και στο τελευταίο παράδειγμα που είναι αυτό της Γαλλίας και αυτό που σας προτείνω ήδη είναι δεδομένης καθυστέρησης τα μέλη του Κοινοβουλίου που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις να το κάνουν μέσω email στην Έρικα, η οποία θα συγκεντρώσει τις ερωτήσεις και θα ε, συγκεντρώσει και τις απαντήσεις. Σας ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρηση και δεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα το κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Για την κατάσταση στη Γαλλία η Γαλλία είναι από τα 10 κράτη που μας παρουσίασαν που έχει ξεπεράσει τους στόχους της Βαρκελόνης. Και ε, για τα νηπιαγωγεία, δηλαδή η ηλικία μετά τα τρία, προνήπιο και νηπιαγωγείο, όπως επίσης και για την πρόσβαση σε δομές για τα παιδιά κάτω από τα τρία. που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποιο είδους επίσημες ε, δομές φροντίδας. Τα 10-15 τελευταία χρόνια το κυρίαρχο στοιχείο ήταν η αύξηση ε, του αριθμού των ε, γυναικών που κρατάνε παιδιά στο σπίτι, οι οποίες όμως είναι εκπαιδευμένες, είναι καταγεγραμμένες ε, στη Μητρώα Προστασίας ε, Μητρότητας και προσφέρουν κατοίκον τις υπηρεσίες τους. Δηλαδή περισσότερο από τις θέσεις ε, στις δομές ήταν η αύξηση αυτή που βοήθησε γιατί αυτές οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μια ιδιαιτερότητα της Γαλλίας που είναι ότι τα παιδιά από τα 2,5 και πριν τα 3 θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο ε, παιδικό σταθμό αλλά είδαμε ότι το 2000 ήταν ένα τρίτο παραπάνω τα παιδιά ε, τα οποία πήγαιναν σε παιδικούς σταθμούς σε σχέση με αυτά που πήγαινε το 2010. Άρα λοιπόν, είπαμε, θα πρέπει να προκρίνουμε την περίπτωση των τριών ετών, να έχουν αυτά σίγουρα θέση και για τα υπόλοιπα παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε. Du développement des services d'accueil, alors il faut d'abord replacer dans, dans le contexte, hein, euh, la France est l'un des pays de για τις χώρες του ΩΣΑ να σας πω πως στην οικογενειακή πολιτική το 4% του ΑΕΠ της Γαλλίας ε, διατίθεται για οικογενειακές πολιτικές ενώ το μέσο του ΩΣΑ είναι το 2,6%. Έχουμε λοιπόν μια πανσπερμία οικογενειακών επιδομάτων αρκετά γενναιόδωρων. Και στα πλαίσια αυτών των μέτρων έχουμε, και αυτό χαρακτηρίζει τη Γαλλία, γιατί είναι αρκετά παρόμοια με τις βόρειες χώρες, επενδύει πολύ στις ε, δομές αυτές για την νηπιακή ηλικία. 1,1% του ΑΕΠ λοιπόν για την ηλικία αυτή σε σύγκριση με το 0,7% που έχουν οι χώρες του ΩΣΑ. Για ποιο λόγο. Είδαμε περνώντας ο καιρός πως αυτό το οποίο καθώς για τις οικογενειακές πολιτικές αρχικά ήταν η προστασία των παιδιών και η βοήθεια στις φτωχές οικογένειες. Και αργότερα, μετά τα τέλη της δεκαετίας του 70 και προς τη δεκαετία του 80, είδαμε τη συμφαλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Παρόλα αυτά, η πολιτική μας κατέχεται από κάποιες αμφισημίες γιατί αφενός θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ελευθερία επιλογής της οικογένειας που είναι μια διπλή ελευθερία, μια ελευθερία επιλογής μεταξύ να εργαστώ ή όχι. Και είναι βεβαίως κυρίως η μητέρα η οποία κάνει αυτή την επιλογή, όχι ο πατέρας και κατόπιν η επιλογή της μεθόδου φύλαξης του παιδιού. Δηλαδή, μία επίσημη μορφή που έχουμε μια σειρά υπηρεσιών που έχουν ε, δημιουργηθεί στη Γαλλία. Ένα άλλο στοιχείο είναι το αντίτιμο που καταβάλουν οι γονείς για να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δομές. Ισχύουν ισοδηματικά κριτήρια τα επιδόματα τα οποία λαμβάνουν έτσι ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εξαρτώνται από το γεγονός πως δεν θα πρέπει το αντίτιμο που καταβάλουν ε, οι γονείς να ξεπερνάει το 12% του οικογενειακού εισοδήματος, το 10% αν είναι δύο τα παιδιά. Υπάρχει λοιπόν μία αμέγιστη τιμολόγηση που χρωματίζει τα όσα μπορούν ε, να προσφέρουν αυτές οι δομές. Και όπως και στο Βέλγιο, η πρόσβαση στο παιδικό σταθμό είναι δωρεάν. Υπάρχουν και άλλα μέτρα οικογενειακής πολιτικής. 16 εβδομάδες γονική, ε, μητρική άδεια, άδεια το και μητρική και 10 μέρες πατρική. Υπάρχει και γονική άδεια που μπορεί να συνδυαστεί με την καταβολή ενός καταποκοπήν επιδόματος και αυτό βέβαια εξαρτάται και από τον αριθμό των παιδιών που έχει κάθε οικογένεια. Μπορεί κανείς να το λαμβάνει για 6 μήνες όταν έχει ένα παιδί, αλλά και για 3 χρόνια όταν κανείς έχει δεύτερο ή τρίτο παιδί. Είχε και περισσότερα. κάτι που συζητούσαμε στο Κοινοβούλιο και που είχε σκοπό να μειώσει το επίδημα αυτό και τη σχετική γονικής άδειας. Είπαμε έξι μήνες, αλλά έξι μήνες με τη χρήση και από τον πατέρα. Έτσι ώστε να έχουμε και μία ποσόστοση για τον πατέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή το 90% όσων χρησιμοποιούν αυτό το επίδημα και την γονική άδεια είναι γυναίκες. Δεν θα πω παραπάνω. Και πέραν αυτού έχουμε και ένα σύστημα εξαιρετικά γενναιόδωρο, ε, είτε φορολογικών ελαφρύνσεων, είτε οικογενειακών επιδομάτων, που συνδέονται με την ανάληψη του κόστους του παιδιού ή του ε, βρεφονιπιακού. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας πως Τα πλεονεκτήματα του γαλλικού συστήματος συνδέονται και με τη δημογραφική εξέλιξη στη χώρα μας, πολύ υψηλή ρυθμή γεννητικότητας και πολύ υψηλή απασχόληση των γυναικών. Από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Έχουμε πολλές δομές που προσφέρονται στη ε, Γαλλία και επίσης με κεντρικό σύστημα διαχειριζόμαστε τα επιδόματα και την χρηματοδότηση αυτών των ε, παιδικών σταθμών και βρυφονιπιακών σταθμών που έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο που διαπραγματεύονται με την τοπική αυτοδιοίκηση για να δούνε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι ανάγκες και μετά διαχειρίζονται το μηχανισμό κατανομής και στις οικογένειες επίπεδο επιδομάτων αλλά και στις δομές που παρέχουν αυτές οι υπηρεσίες. Ένα λεπτό για να σας πω πώς αυτή τη στιγμή ακολουθούμε μια προσπάθεια να αυξήσουμε τις θέσεις που προσφέρονται. Πρόσφατα ψηφίσαμε μια μείωση των δαπανών, περικοπή δηλαδή των επιδομάτων, των χρηματικών επιδομάτων, αλλά ως αντίβαρο επιβεβαιώσαμε τη βούλησή μας να αυξήσουμε τον αριθμό των θέσεων. Από τις 275.000 γιατί είμαστε λίγο κάτω από αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θέλουμε 400.000 τελικά για να καλύψουμε όλες τις οικογένειες και βεβαίως έχουμε τη βούληση να αυξήσουμε και την δυνατότητα πρόσβασης των φτωχών οικογενειών ή των μειονοτήτων. και κυρίως γιατί προσφέρονται πλέον εκτήματα για την ένταξη στην κοινωνική αυτών των παιδιών και για το μέλλον του στο σχολικό. Dans le sens, je crois y a une euh, avec... Αυτό λοιπόν και για να μην υπάρχει σύγχυση Πιστεύω και εγώ τα ίδια με τους προλανήσαντες, οι μελέτες όντως επιβεβαιώνουν πως το να έχει κανείς πρόσβαση σε τέτοιου είδους επίσημες δομές με έρημνας η φροντίδας προσχολικής αγωγής έχει θετικό αντίκτυπο στην γνωστική εξέλιξη των παιδιών και κυρίως για τις οικογένειες που μειονεκτούν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονές μας για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ακρόση. Ευχαριστή πρόεδρος και τους ε, διερμηνείς, όλους ιδιαίτερος, που έπαιξαν στην παράταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές που έμειναν.